Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε αυτή τη συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θέμα. Πάντα θα είναι επίκαιρο τους επόμενους μήνες, κυρίως όταν μιλάμε για τις ε, νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Το ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη για εσά τη ημερήσια τη συνεδρία σα Έχουμε μια μικρή αλλαγή. Αντί συζητήσουμε από 9 μέχρι 11 και 30, οι συζητήσει θα λάβουν χώρα από 9 μέχρι 11, διότι στι 11 θα γίνει η ειδική συζήτηση για την απαλλαγή του Συμβουλίου ε, και γι' αυτό όλοι θα πρέπει να περιοριστούν όσον αφορά τις συνεισφορές τους. Να μην μιλήσουν πιο γρήγορα, αλλά να είναι συντομότεροι, συνοπτικότεροι στα σχόλιά τους. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπάρτ Στάς. Ε, Μπάρτ, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι, εξετάζουμε ένα σημαντικότατο θέμα σήμερα – Οι λόγοι πίσω από αυτή την ακρόαση ξεκίνησαν από έναν χρόνο περίπου, όταν διαπιστώσαμε μέσω του τύπου κυρίως ότι κάποια οικολογική μαφία είχε διεισδύσει στην, στον τομέα των ανεωσίμων πηγών ενεργείας στην Ιταλία και στο άρθρο αυτό της εφημερίδας αναφερθήκαν διάφορες επιχειρήσεις της αστυνομίας που η αστυνομία εξέταζε με κάθε σοβαρότητα την εγκληματικότητα, την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε διάφορους τίτλους όπως ε, πήρε ο άνεμος» Φερρυπίν. Ε, εξαφανιζόταν χρήματα, όχι μόνο ευρωπαϊκά, αλλά και ε, ιταλικά, λόγω ατασταλιών, στον τομέα της αιωλικής ενέργειας. Ε, γνωρίζουμε ότι αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Ισπανία, Ρουμανία, Γαλλία, ε, στην Κορσική, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Περνάμε δύσκολες εποχές, έχουμε οικονομική και ε, δημοσιονομική κρίση, χρηματοπιστική κρίση. Πρέπει σαν Ευρωπαίοι να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα δημόσια χρήματα γίνονται συζητήσεις για το μέγεθος του ευρωπαϊκού προπολογισμού και πολύ συχνά αναφέρεται ότι ίσως δεν θα έπρεπε να τίθενται περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι, θα έπρεπε να δούμε όχι την ποσότητα αλλά την ποιότητα, το πώς απορροφώνται τα χρήματα και το σημερινό εγχείρημα αυτό το σκοπό έχει. Ε, θέλουμε να δούμε πώς κάποια ποσά από τα ευρωπαϊκά χρήματα ε, αποτελούν δικείμενο διαχείρισης, πώς τα χειριζόμαστε, ποιοι είναι εκείνοι που πραγματικά ωφελούνται από τις επιδοτήσεις ε, και αν, αν, ωφελούνται, αν με, με το σωστό τρόπο. Θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα λεπτομερέστερα. Έχουμε ένα πάνελ με πάρα πολλούς ε, καλούς επαΐοντες και προσβλέπω στο να ακούσω αυτά που έχουν να μας πούν Οπότε εμείς ελπίζουμε σαν Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού να μπορούμε να συναγάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα για το μέλλον, κυρίως όσον αφορά την απαλλαγή που θα συζητήσουμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Μπάρτ. Με τα χαράς, στον κύριο Φαζάκας να δώσω το λόγο, έναν τους προκατόχους μου σε αυτή τη θέση και μέλος τώρα του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συμμετέχοντες, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το, την Επιτροπή και ιδίω τον εισηγητή Μπάτ Στάς που οργάνωσε αυτήν την συνεδρίαση διότι ε, σαν εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω αυτή την ε, ομιλία για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας και καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μιλντερ σαν πρόεδρο αυτής της Επιτροπής διότι είμαι προκάτοχός σας αυτή τη θέση και ε, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθεί κανείς την ποιότητα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είμαι ένας φίλος σας και είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο έχετε τις αναγκαίες γνώσεις αλλά ε, και ε, την, τις ικανότητες για να καλύψετε τη θέση σας και γι' αυτό ε, σας παρακαλώ να δεχθείτε ε, τις διαβεβαιώσεις μου ε, για την στήριξη που θα σας παρέχω. Η σημερινή κρίση όμως αντιπροσωπεύει πολλές προκλήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να δούμε πώς θα επιληθούν οι λύσεις αυτές διότι όπως γνωρίζετε ε, το ε, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανεξάρτητο σώμα και ε, αποτελεί έναν στυλοβάτη που στηρίζει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες προτάσεις σχετικά με τις δαπάνες και, και ε, εμείς δεν ελέγχουμε ε, τις ε, πολιτικές αποφάσεις αλλά μόνο ο πώς έχουν δαπανηθεί τα χρήματα διότι ο ρόλος μας είναι να γίνεται σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού με τη διπλή του όμως θέση το Κοινοβούλιο σαν συνομοθέτη της και ελεγκτής μπορεί να ελέγξει τις δαπάνες αυτές και γι' αυτό ε, η εντολή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πολύ ευρεία ε, ε, και καλύπτουμε τη συμμόρφωση από πολλές οπτικές γωνίες και δεν εκφράζουμε τη δική μας γνώμη αναφερόμαστε στη συμμόρφωση στα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία χρειάζονται για να υπάρχει σωστή χρήση των δημοσίων πόρων. Γι' αυτό και η σωστή αξιοποίηση των πόρων είναι μια νομική δέσμευση και ε, πρέπει ε, να παρουσιάζουμε μία ε, γνωμοδότηση κατόπιν του ελέγχου και εφόσον έχουμε ελέγξει όλες τις πτυχές Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Ε, εάν όμως σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει όπως στον τομέα της συνοχής, το επίπεδο ε, των ε, παρατυπιών δεν θεωρείται από το από το ελεγκτικό συνέδριο σαν ε, ε, ε, διαφθορά αλλά απλούστατα θεωρούμε ότι υπάρχουν παρατυπίες οι οποίες αναφέρονται εις τα συμπεράσματα κατόπιν της εκθέσεως η οποία υιοθετήθηκε πέρυσι και γι' αυτό παρουσιάζουμε πόσο πραγματικά δαπανήθηκαν οι πόροι και διατυπώνουμε προτάσεις σύμφωνα με τις αρχές οικονομίας αποτελεσματικό και αποτελεσματικότητος. Ε, πέρυσι είχαμε υιοθετήσει 14 ειδικέ εκθέσεις που αναφέρονται εις τους πόρους και στον τομέα της ενεργείας και των υπηρεσιών υπήρχαν διάφορα προγράμματα εν εξελίξη όπως είναι ε, το κλείσιμο πυρνικών σταθμών ή ε, αναδιαμόρφωση του οδικού συστήματος και άλλα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. Τέλος, οι προτάσεις για αναθεωρημένες ρυθμίσεις ε, με ε, οικονομικές επιπτώσεις επίσης πρέπει να τονιστούν και γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναφερθεί στις βελτιώσεις σε διάφορους τομείς όπου που ε, μπορεί να υπάρξει μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Το στόχος του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είναι να υποδείξει πού μπορούμε να δαπανίσουμε περισσότερα αλλά καλύτερα και ε, οποιαδήποτε δαπάνη ε, δεν επαρκεί. Πρέπει να υπάρχει μία ποιοτική και ποσοτική διάσταση και η αφομοίωση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για εύκολη δαπάνη. Τώρα, σχετικά με τις ερωτήσεις που είχατε κάνει σχετικά με τους αποδέκτες, ε, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν πραγματικά ωφέλη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να σας τονίσω ότι άλλο είναι να είναι κανείς αποδέκτης και άλλο να είναι ο τελικά ωφελημένος ε, διότι στον ε, τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προβλέπονται το μίσο που υπάρχει συγχρηματοδότηση όπως η συνοχή και άλλες και υπάρχει μία αμοιβαία αλληλεπίδραση. Οπότε οι τελικοί αποδέκτες δεν ε, χρηματοδοτούνται ε, επιπρόσθετα υποχρεωτικά ε, λόγω της επεμβάσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι χρειάζεται και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και η εθνική συμμετοχή και πρέπει να έχουν επιλεχθεί και τα προγράμματα τα οποία θα, θα συγχρηματοδοτηθούν υπάρχουν ορισμένοι τομείς πιο ευαίσθητοι όπως είναι η έρευνα αλλά ή σε την γεωργία, στην αλληλεία, το, η ε, καθημερινή διαχείριση των προγραμμάτων αναλαμβάνεται από τα κράτη-μέλη διότι υπάρχει μία μοιρασμένη διαχείριση και αυτοί αναλαμβάνουν την ε, αποστολή των πόρων στους τελικούς αποδέκτες. Είναι δηλαδή διάφοροι τομείς στους οποίους μόνο οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση και βλέπουμε ότι στην πολιτική συνοχής ε, υπάρχει μία πλήρης χρηματοδότησης πολλές φορές από τους εθνικούς πόρους παρόλο που δεν υπάρχει λόγος κανείς να θεωρήσει ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων. Αλλά θα λέγαμε ότι συμπλέουν ο ευρωπαϊκός προπολογισμός και η εθνική οι πόροι διότι πρέπει να έχουμε υπόψη ε, ε, ποιοι είναι επιλέξιμοι και ε, ποιοι όχι ιδίω όταν πρόκειται για δημόσιους, δημόσιες προμήθειες και ο τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα γίνουν νομότυπα είναι να ελέγχουμε το τα μέτρα για να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε ε, να ε, βελτιώνουμε συνέχεια τον έλεγχο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πρέπει να υπάρξουν και αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεται το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο με συγχωρείτε, την ε, σημασία της αξιολογήσεως των δημοσίων πολιτικών και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ εις ε, την εγκύκλειό μας ε, διότι το, αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το πόσο ξοδεύονται τα χρήματα αλλά ποιο είναι το περιεχόμενο των πολιτικών και τέτοιες τάσεις πρέπει να αξιοποιηθούν στις επόμενες στην επόμενη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με ε, την πολιτική συνοχής ε, μετά το 2013 και το σχετικό κανονισμό κατά τρόπον ώστε να εστιαστούμε ε, στα αποτελέσματα και εις ε, και να μην περιοριστούμε στην τακτικότητα ε, της ε, χρηματοδοτήσεως. Ε, και καταλήγοντας επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι συνάδελφοί μου στο ελεκτικό συνέδριο και εγώ είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται μία ολοκληρωμένη προσπάθεια από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συνεργασία μας με όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαιτέρως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει αποτελεσματικότητα προς όφελος των ε, αποδεκτών, των Ευρωπαίων φορολογουμένων και του συνόλου Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια που είπατε στην εισαγωγή σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σλότερς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, um, Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής στη συνάντηση αυτή. Uh, Αυτό που θέλω να κάνω στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για την παρουσίασή μου είναι να σας προσανατολίσω εν συντομία μέσω μιας επισκοπήσεως των συγχρηματοδοτωμένων προγραμμάτων στα δομέα ανανεωσίμων πηγών ενεργείας και αποδοτικότητας ενέργειας στην Ιταλία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην Νότια Ιταλία και θέτοντας και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να δούμε πού στέκεται η Νότια Ιταλία ε, σε σχέση με την Ιταλία και σε σχέση με την Ευρώπη. Μπορεί να ξεκινήσουν οι διαφάνειες.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 Ωραία, έχουμε την εικόνα, έχουμε τις διαφάνειες. Μπορείτε να πάτε πιο πέρα σε μια, στην διαφάνεια. Στο πρώτο διάγραμμα που σας παρουσιάζω Βλέπετε τις δαπάνες που από 5 Οκτωβρίου του 2011 έχουν πραγματοποιηθεί από τις βασικές δικαιούχες χώρες των διεθνωτικών ταμείων σε εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπετε οι δαπάνε όσον αφορά τι ανώνυμε πηγέ ενέργεια και την αποδοτικότητα τη ενέργεια, διότι αυτό αντιπροσωπεύεται εδώ. Στην Ιταλία σχετικούς αριθμούς είναι αρκετά υψηλό το ποσό σε άλλες χώρες. Η Ιταλία μέχρι τώρα έχει πάει περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις δύο κατηγορίες των δαπανών. Και νούμερο δύο, αν μπορούμε να το πούμε στον κατάλογο, είναι η Ισπανία, η Γαλλία, 150.000 περίπου λέει ο σε σχέση με άλλε χώρε, λοιπόν, όσον αφορά την αποδοτικότητα τη ενέργεια και ανανεώσιμε πηγέ ενεργεία, βλέπετε ότι τα ποσά είναι πάρα πολύ ψηλά στην Ιταλία. Να τονίσω επίση ότι όσον αφορά το Γενικό Χαρτοφυλάκιο των Θετικών Ταμείων για την Ιταλία στην περίοδο 2007-2013, είναι σχετικά μικρά ποσά αυτά. Λάβετε υπόψη το συνολικέ δαπάνε για την Ιταλία των προγραμμάτων που είναι τη τάξη των 55 με 60 δι. Οπότε 300.000 που βλέπετε εδώ, λέει ο είναι σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. 0,5% περίπου αντιπροσωπεύει, άρα βλέπουμε σχετικά το σχετικό βάρος ε, του προγράμματος αυτού στα προγράμματα που χρηματοδοτούν στην Ιταλία. Εδώ βλέπετε τις ίδιες πληροφορίες με διαφορετικό γράφημα, πιο εύληπτο γράφημα. Πάμε τώρα στο τι έχει κατασταθεί μέχρι τώρα όσον αφορά το δυναμικό ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στην Ιταλία για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πιο συγκεκριμένα. Βλέπετε εδώ μερικά στοιχεία. Στην πρώτη στήλη βλέπετε τον αριθμό για το συνολικό δυναμικό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διάφορες χώρες και βλέπετε στη δεύτερη στήλη το ποσοστό ανανεωσίμων πηγών ενεργείας όσον αφορά το συνολικό δυναμικό και ακολουθείτε το συνολικό δυναμικό ανανεωσίμων πηγών ενεργείας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ε, βλέπετε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν πάρουμε την τελευταία στήλη, που είναι ο δείκτης λίγο πολύ, διείσδυσης ανανοσίμων στη χώρα, βλέπετε το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, που είναι της τάξης των 470 και η Ιταλία δεν είναι μακριά, από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, όπως θα αναμενόταν χώρες όπως είναι η Αυστρία και η Σουηδία, τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Έχουν πολύ ψηλότερο μερίδιο ανανοσίμων πηγών ενεργείας στην γενική παραγωγή ενέργειας, συνολική παραγωγή ενέργειας. Τώρα πάμε στην Ιταλία και τους τρεις τομείς εντός Ιταλίας, τις τρεις περιοχές. Βλέπετε ότι στο Νότο, αν πάρουμε το Μεσοτζόρνο, την Νότια Ιταλία, εκεί που είναι φωτισμένη η γραμμή, ξεκίνησε το 2000 με αγκατεστημένες πηγές ανοσίμων πηγών μόνο τριών ε, εκατομμυρίων, γρήγορα το 2009 και πήγε το 2010 σε 10,5 χιλιάδες μεγαβάτ εγκατεστημένα. Οπότε το γενικό ποσοστό ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές στη Νότια Ιταλία, στο Μεζοτζόρνο, αυξήθηκε από 12 που ήταν αρχικά της 100, από 12% πήγε στο 32%. Οπότε είδαμε σημαντική προσπάθεια καλύψεως των καθυστερήσεων, διότι το 2000 η διείσδυση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στην Νότια Ιταλία ήταν πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ιταλίας. Και το βλέπετε αυτό σε γραφική παράσταση στην επόμενη διαφάνεια, όπου βλέπετε ποιες είναι οι τάσεις για τις ανανεώσιμες στο Μεσοτζόρνο. Βλέπετε την πράσινη γραμμή που ανέρχεται με μεγαλύτερους ρυθμούς, υψηλότερους ρυθμούς από ότι το κέντρο, η κεντρική Ιταλία και η βόρεια Ιταλία. Τώρα όσον αφορά τη σύνθεση του εγκατεστημένου δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές στην Ιταλία βλέπουμε και κάποιες διαφορές στις διάφορες περιοχές. Στο βορρά η περισσότερη ενέργεια, 80%, προέρχεται από υδροηλεκτρική ενέργεια και γεωθερμική ενέργεια. Βλέπετε στην πρώτη γραμμή της διαφάνειας. Στο κέντρο της Ιταλίας περίπου 70% προέρχεται από αυτές τις δύο πηγές αλλά περισσότερο ποσοστό από φωτοβολταϊκή ενέργεια. Μεγαλύτερο δυναμικό φωτοβολταϊκό από ότι στο βορρά. Στο νότο η, υδροδυναμ... υδρο... η παραγωγή από νερό είναι μικρότερη, αλλά η ολική είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι κοντά στο 50% από το συνολικό δυναμικό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νότο. Αυτά είναι στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί βάσει των δικών μας εκθέσεων και βάσει εκθέσεων των Ιταλικών αρχών και Ιταλικών εταιριών. Τώρα, στρεφόμενοι στη, στη Κελία και κάποιες άλλες περιοχές της Ιταλίας, πιο συγκεκριμένα, η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει τι είναι εγκατεστημένο, τι έχει εγκατασταθεί, τι έχει συγχρηματοδοτηθεί και τι έχει εγκατασταθεί στη Σικελία. Ε, το ROP είναι τα περιφερεια... ROP, Regional Operational Programs, τα περιφερειακά προγράμματα στην Ιταλία. Βλέπετε το συγχρηματοδοτούμενο δυναμικό που έχει εγκατασταθεί απαρτίζεται κυρίως από αιωλική ενέργεια. Δεν μας εκπλήσει αυτό, είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια ότι στην Νότια Ιταλία είδαμε ότι κυρίως η ολική ενέργεια είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναλλακτικών μορφών ενέργειας. Και η τρίτη στήλη μας ενδιαφέρει που δίνει το συνολικό δυναμικό που έχει εγκατασταθεί στη Σικελία κατά πηγή και βλέπετε υπολογίζοντας το ποσοστό του συγχρηματοδοτούμενου δυναμικού και του συνολικού εγκατεστημένου δυναμικού βλέπετε ότι το μερίδιο της του συγχρηματοδούμενου δυναμικού είναι αρκετά χαμηλό. Για όλες τις ανανεώσιμες πηγές μαζί είναι περίπου 16% και στο νεολικό τομέα είναι ακόμα λιγότερο από το 16%. Οπότε η επιρροή της χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή Ένωση στις στην εναλλακτική ενέργεια, κυρίως από φωτοβολταϊκές πηγές περισσότερο από τους άλλους δύο τομείς, αιωλική ενέργεια και βιομάζα. Η βιομάζα είναι σχεδόν αμεληταία. Ο υλικό τομέα είναι ο σημαντικό από πλευρά κοινοτική συγχρηματοδότηση. Δεύτερη σημασία. Πάμε σε επόμενε δύο διαφάνειε. Βλέπετε για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην Ιταλία τις παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα που χρηματοδοτούνται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ο αριθμός των προγραμμάτων, το κόστος αυτών και τις ε, πληρωμές τις σχετικές. Πάμε στην άλλη διαφάνεια. Ε, και σύμφωνα με κάθε περιοχή τι, γίνεται και ανάλογα με κάθε πρόγραμμα τι γίνεται. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, Βλέπετε, αιωλική ενέργεια τώρα είναι σχετικά λιγότερο σημαντική αν δούμε όλα τα προγράμματα που είναι 1,4 δις που έχουν προγραμματιστεί στην προτελευταία στήλη πριν από τα ποσοστά το βλέπετε αυτό για ολική ενέργεια είμαστε στα 50 εκατομμύρια και ηλιακή, φωτοβολταϊκή είναι 245. Η πιο σημαντική κατηγορία είναι ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή όχι παραγωγή, αλλά αποδοτικότητα. Κοντά στα 600 εκατομμύρια. Οπότε βλέπουμε τη σχετική σημασία των διαφόρων τομέων ανανοσίμων πηγών ενεργείας στις διάφορες περιοχές της Νότιας Ιταλίας. η παρούσα κατάσταση, ζητώ συγγνώμη, διότι είναι στοιχεία αυτά που ελήφθησαν, είναι στοιχεία μέχρι 31 2010, είναι τα πιο αξιόπιστα στοιχεία, έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία, αλλά αυτά είναι τα πιστοποιημένα αξιόπιστα στοιχεία. Βλέπουμε τη γενική κατάσταση των πληρωμών, τα 300 εκατομμύρια που ήδη προαναφέραμε στην ε, πρώτη διαφάνεια και βλέπετε πώς διαχωρίζονται οι διάφορες περιοχές καθέτως και τομεακά όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οριζόντια, κυρίως η ηλιακή έχει πάει τα περισσότερα χρήματα και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Όσον αφορά τις πραγματοποιηθήσεις δαπάνες, είμαστε ακόμα στο μηδέν όσον αφορά την αιωλική ενέργεια που συγχρηματοδοτείται στην παρούσα ε, προγραμματική περίοδο. Οι επόμενες δύο διαφάνειες δείχνουν τρόπο, μάλλον είδος γραφήματος, την κατάσταση. Ήθελα να υπογραμμίσω στην παρουσίασή μου ότι πράγματι χρηματοδοτούμε με σημαντικά ποσά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία και κυρίως στην Νότια Ιταλία. Όμως, εν συγκρίση με την διαθέσιμη ιταλική χρηματοδότηση για τον τομέα, καθαρά ιταλική, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι σχετικά ίσονο σημασία. Καλύπτουν λιγότερο το 16% του γενικού δυναμικού που έχει εγκατασταθεί και καθίσταται. Όσον αφορά το διαχωρισμό μεταξύ τομέων, αυτό που διαφαίνεται σαφώς είναι ότι μέχρι τώρα έχουμε χρηματοδοτήσει πάρα πολύ λίγο την αιωλική ενέργεια και ο σχεδιασμός για την υπόλοιπη τετραετία της προγραμματικής περίοδου δείχνει ότι θα αυξηθεί αυτό, αλλά όχι πάρα πολύ, διότι τα προγράμματα της Νοτιού Ιταλίας εστιάζονται τώρα σαφώς στην ηλιακή ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και εκεί δίνουμε τη μεγαλύτερη σημασία στον αφορά τα κίνητρα που δίνουμε. Θα ήθελα να δείξω με μια τελική διαφάνεια αυτά που έλεγε ο κ. Φαζάκας. Έλεγχος, το πλαίσιο ελέγχου ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και στην Ιταλία, όσον αφορά την κοινή διαχείριση. Για κάθε πρόγραμμα έχουμε τρεις αρχές, διαχειριστική αρχή. Αρχή πιστοποίησης που πιστοποιεί τις δαπάνες και ελεγκτική αρχή που ελέγχει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα στην περιοχή. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο επίπεδα ελέγχων. Η διαχειριστική αρχή αυτή η ίδια πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη και τη σωστή εκτέλεση κάθε προγράμματος που συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος για το οποίο φέρει ευθύνη. Η πιστοποιού αρχή πραγματοποιεί δεύτερο έλεγχο όταν μας δηλώνει τις πληρωμές, μας πιστοποιεί ότι είναι νόμιμες και κανονικές πληρωμές και η ελεκτική αρχή, η οποία αποτελεί τμήμα επίσης της ελεγκτικής δομής του προγράμματος, η αρχή ελέγχου ελέγχει και τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης. Και επιπλέον υπάρχουν και υπηρεσίες ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG Regio ε, και άλλοι φορείς ελέγχου που ελέγχουν την ελεγκτική αρχή. Και κάνουν και επισκέψεις επιτόπου για να δουν ε, πώς πηγαίνουν τα διάφορα προγράμματα και πώς γίνονται κινήσει σε επίπεδο πιστοποιούσας αρχής και διαχειριστική αρχής. Θα ήθελα να σταματήσω κάπου εδώ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ νέου που με καλέσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας και ελπίζω ότι είμαστε έτοιμοι μάλλον θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε για θέματα που σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολίνο Παραγκόνα από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης είμαστε η αρμόδια αρχή όσον αφορά τις επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε σχέση με το πλαίσιο που μας, ε, μόλις σας εξέθεσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμείς από πλευρά Ιταλίας θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς διαρθρώνονται οι επενδύσεις ε, σε σχέση με το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ενέργεια και το περιβάλλον με τη χρήση βιώσιμων πόρων για την ανάπτυξη και έπειτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της, ε, της αρμόδιας περιφερειακής αρχής της ΕΚΕ για να δώσει κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση. Στόχοι του Εθνικού Πλαισίου ανάπτυξη είναι η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω τη ανάπτυξη παραγωγικών θηγατρικών σε σχέση με την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργεια Κάποιε πληροφορίε ήδη σα δόθηκαν από την Κομισιόν όσον αφορά τα προγράμματα με πιο ε, τελευταίες πληροφορίες είναι στοιχεία της 31ης Αυγούστου 2010 αλλά έκτοτε υπάρχει πρόοδος σε σχέση με τα στοιχεία που είχατε παλιότερα. Χωρίς να μπούμε όμως σε λεπτομέρειες και σε αριθμητικά στοιχεία, θα έλεγα καταρχήν πως οι πόροι που έχουν ε, προβλεφθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο και προβλέπονται στο πλαίσιο 2007-2013 ανέρχονται στα 3 δις όσον αφορά το στόχο σύγκλησης και ένα δις όσον αφορά το στόχο ανταγωνιστικό, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και ε, συντονισμός. Ε, τώρα, σε σχέση με όλα αυτά, πού αναφερόμαστε όσον αφορά τις ε, στρατηγικές επιλογές. Καταρχήν, στήριξη όσον αφορά τη δημιουργία και την ε, παγίωση παραγωγικών θηγατρικών που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ε, τις οικονομικές ε, παρεμβάσεις που προέρχονται για, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλη μια στρατηγική επιλογή είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σε θέματα ανανεώσιμης ε, ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Άλλη μια επιλογή είναι η ενδυνάμωση του δικτύου διανομής και τέλος Υπάρχει και ο στόχο τη διάδοση γνώσεων και τεχνογνωσία όσον αφορά τι καλύτερε πρακτικέ για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της στρατηγικής επιλογής ήταν και η δημιουργία όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της σύγκλησης πέρα από τις επενδύσεις σε μεμονωμένα προγράμματα και ένα διαπεριφερειακό πρόγραμμα το οποίο είχε στόχο να στηρίξει τις επιλογές παρέμβασης ε, υπερεθνικής ε, αξίας για να ενισχύσει όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες ε, του τομέα. Αυτές ήταν οι στρατηγικές επιλογές που αποτελούν την βάση αυτής της δραστηριότητας. Η κατάσταση των επενδύσεων τώρα, πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία μπορεί να έχετε, στη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή είναι κάπως παλιότερα όσον αφορά την περίοδο 2007-2013 όπου οι εθνικές αρχές έχουν προσπαθήσει να ε, εξασφαλίσουν ορίζοντας ε, στόχους ώστε αν δεν επιτευχθούν αυτοί μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις απέναντι προς τις αρχές οι οποίες είχαν κληθεί να διαχειριστούν τα προγράμματα. Και αυτή η εξασφάλιση έδωσε σε καλά αποτελέσματα γιατί στις 31 Αυγούστου, αν και έχουμε καθυστέρηση, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ε, σε προηγούμενες αντίστοιχες ε, περιπτώσεις. Για να σας δώσω μόνο κάποια στοιχεία, ο αριθμός των προγραμμάτων που έλαβε χρηματοδότηση και που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχει περάσει σε πάνω από 2.000. Νομίζω πως την τελευταία φορά η ενημέρωση της Κομισιόν μιλούσε για τα μισά ε, προγράμματα από αυτά. Τώρα, τι αφορούν αυτά τα προγράμματα. Καταρχήν, όπως είπα ήδη, μιλάμε για ενεργειακή επάρκεια, παρεμβάσεις ε, σε ε, δημιουργία δημόσιας ε, ε, ηλεκτροδότησης, ε, διανομής όσον αφορά την ανανεώσιμη, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η υδροηλεκτρική, αιωλική και σύνδεση αυτών με τα δίκτυα θέρμανσης και άλλες εγκαταστάσεις που αφορούν την έναρξη και την ενίσχυση στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αστικές περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την Σικελία. Ε, τώρα, πώς έγινε η επιλογή των προγραμμάτων. Ε, καταρχήν, ε, όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε εσωτερική, στην εσωτερική αγορά, τηρήσαμε τις σχετικές αρχές, αλλά και τις αρχές που καθορίζονται στα σχετικά προγράμματα και στους σχετικούς κανονισμούς. Δηλαδή, τα κριτήρια ποια είναι. Συνοχή με το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε περιφερειακό επίπεδο, σεβασμός ε, της ε, παραγωγής η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ε, της χρήσης της ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εγγύηση της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης στις τοπικές ε, επιχειρήσεις. Όλα αυτά βεβαίως υλοποιούνται χρησιμοποιώντας τις ε, διαδικασίες που προβλέπονται από τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των μεμονωμένων προγραμμάτων που ε, υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που διαρκώς ε, υποβάλλονται σε ελέγχους τόσο από την εσωτερική διαχείριση όσο και από την κοινότητα. γίνονται έλεγχοι από το ελεγκτικό συνέδριο και από την DG Radio. Πιστεύω πως σε αυτή τη φάση θα ήταν καλό η περιφέρεια της Σικελίας να δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επιτόπου. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Τζανλούκα Γαλάτη. Είμαι διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας για την περιφέρεια της Σικελίας. Ήθελα να προσθέσω, μάλλον επιβεβαιώσω για την Σικελία αυτά που είπε ο προηγούμενος ε, και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην περιοχή της Σικελίας. Σύμφωνα με το ενεργειακό μας πρόγραμμα σχέδιο έχουμε να διαμορφώσει την χρήση των πόρων 2007-2013 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και όπως αναφέρθηκε και παρουσιάστηκε στις διαφάνειες που είδατε, υπάρχει από την πλευρά μας αλλαγή πορείας. Δηλαδή, προσπαθούμε να αποθαρρύνουμε εκείνους που έχουν τις μεγάλες καταστάσεις, ε, ε, τις ολικές εγκαταστάσεις, είναι η τέταρτη σε παραγωγή ενέργειας από ολική ενέργεια, η περιοχή μας, και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση των πόρων των ευρωπαϊκών για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και, για την, και τη χρήση από βιομάζα, κυρίως με εγκαταστάσεις μέσης και μικρής, μικρού μεγέθους. Και θέλουμε να εκδοθούν περισσότερο οι παρεμβάσεις αυτές στην όλη περιοχή. Όλα αυτά προσπαθώντας, αν και είναι περίπλοκο να πετύχουμε ε, τους στόχους του burden sharing, που συμμετέχει και η Ιταλία και η Σικελία και επειδή είναι περίπλοκο χρειάζονται πάρα πολλές παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε στο βαθμό του δυνατού την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές ενέργειας αλλά επαναλαμβάνω προσπαθώντας να πετύχουμε το στίχημά μας δηλαδή να ευνοήσουμε μεγαλύτερη διάδοση στην περιοχή Μικρότερες εγκαταστάσεις, περισσότερη φωτοβολταϊκή ενέργεια μέσου μεγέθους και μικρές εγκαταστάσεις ε, παραγωγής ενέργειας από τη βιομάζα. Όλα αυτά ουσιαστικά τα κάνουμε μέσω δύο βασικών παρεμβάσεων που ανέφερε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Δηλαδή ε, παραγωγή, τον τομέα της παραγωγής και την ενεργειακή απόδοση. Αυτά τα μέτρα στρέφονται κυρίως προς το δημόσιο τομέα, διότι η κατάσταση όσον αφορά ενεργειακή απόδοση είναι πραγματική πρόκληση που πρέπει να επιτευχθεί. Οι στόχοι του burden sharing να επιτευχθούν. Έχουμε πρόθεση να διαθέσουμε μεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών πόρων στο θέμα και στα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και μέσα τυπικά κοινοτικά όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Σύμφωνο των Νησιών για να ε, μπορέσουμε να κάνουμε συμμετάσχη ο δημόσιος τομέας για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους στη Σικέλια και να χρησιμοποιήσουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, επαρκή προσοχή και συνομιλούμε με το δημόσιο τομέα και με τις μεγάλες επιχειρήσεις από την άλλη που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας. Δίνω το λόγο στον κύριο Μαρίνο. Εμείς κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά το 2007-2013. Οπότε θα μιλήσει ο επόμενος ομιλητής για το θέμα. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, ο πρόεδρος δίνει το λόγο στους ομιλητές και όχι τα μέλη της αντιπροσωπείας. Πόσοι ομιλητές ακολουθούν από την Ιταλία, διότι είναι πάντα, με εκπλήσει ότι πάντα υπάρχει ένα σύστημα αλληλουχίας. Πόσοι ομιλητές θα μιλήσουν ακόμα από την Ιταλία. Πόσους ακόμα έχουμε να μιλήσουν. Ένας. Δεν έχουμε παραπάνω. Πόσο χρόνο θέλετε να μιλήσετε προτίθεστε να μιλήσετε. Εστέ σύντομο παρακαλώ. Δέκα λεπτά λέει ο μιλητή. Και λιγότερο. Δέκα λεπτά είναι πάρα πολλά. Πέντε λεπτά λέει ο πρόεδρο. Πέντε συμφωνεί και ο εμπειρογνώμο. συγγνώμη από εσά κύριε πρόεδρε. Δεν θέλαμε να παραβούμε τους κανόνες. Ήταν η πρώτη μου παρουσία εδώ, δεν είχα εμπειρία και γι' αυτό το έκανα. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε μια πολύ σύντομη παρέμβαση. Ακούσατε λοιπόν τον Δ. Καλάτε για το πώς η Σικελία, η κυβέρνηση της Σικελίας θέλει να αναπτύξει και να υποστηρίξει τον τομέα των ανεσίμων πηγών ενέργειας. Και έχουμε αναλάβει και άλλη δέσμευση παράλληλα και καταβάλουμε προσπάθειες για να χρησιμοποιήσουμε όλα τα τα μέτρα που προέρχονται από την εθνική και περιφερειακή νομοθεσία για να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των πόρων και να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία ή διάφορα κλιματικά φαινόμενα. Θα ήθελα να πω συντομία ότι φέτος πρότεινα και πέτυχα υπογραφή πρωτοκόλλου με την οικονομική αστυνομία, με τη φορολογική αστυνομία στην Ιταλία. που εποπτεύει αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικές σε αυτό το τομέα. Και εγκληματικότητα, ε, ο εγκληματικός τομέας ίσως να θέλει να κινηθεί και σε αυτόν όπως άλλους. Με το πρωτόκολλο αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε κάθε εξουσία, όλες τις άδειες για την υλοποίηση εγκαταστάσεων, να τις δίνουμε σε αυτή την ε, οικονομική αστυνομία για όλες τις δραστηριότητε της κοινοφελής και του δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε η οικονομική αυτή αστυνομία να κάνει διακριβώσεις κατά πόσο γίνονται σωστά τις διαδικασίες να κάνει συνεχώς εποπτεία και να επαληθεύει πώς λειτουργούν όλοι οι φορείς στον τομέα. Για να καταστήλουμε ή δυνατόν, να αποφύγουμε και να καταστήλουμε τη διείσδυση του κλιματικού τομέα και τη αστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το πρώτο εργαλείο. Και έχουμε και ένα άλλο πρωτόκολλο που υπέγραψα με το Υπουργείο, το Υπουργό Συντερικών, τον κύριο Μαρόνι, και με, τους, με τον νομάρχη της Ιταλίας πριν ήμουν νομάρχης στο Παλέρμο, Σικελία. Λοιπόν, υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το οποίο πριν δοθεί άδεια για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων να γίνονται εξακριβώσεις, να δούμε αυτοί που ζητούν την άδεια τι ποιοι είναι, να γίνει επαλήθευση. Τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες επίσης των εδαφών επί των οποίων κατασκευάζονται οι καταστάσεις. Ποιοι είναι αυτοί. και εκείνοι που αγοράζουν τι εγκαταστάσει ποιοι είναι. Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στι προσπάθειε. Είναι πολύ καλά εργαλεία, αποτελεσματικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών. Αυτό κάνει συγκελία. και θα ήταν καλό να γίνεται παντού, για ένα λόγο και μόνο, κυρίες και κύριοι. Το οργανωμένο έγκλημα δεν επενδύει σε συγκεκριμένε περιοχές και μόνο. Έχει πολλά χρήματα. Και επενδύει εκεί που έχει τα μεγαλύτερα κέρδη επενδύοντας τα χρήματα. Εκτός κράτους, εκτός περιφ... και εκτός... βγαίνει εκτός συνόρων συγκεκριμένων. Μια τέτοια μεθολογία, αν εφαρμόζεται, θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Διότι δεν αποκλείεται κάποιες εγκληματικές οργανώσεις από κάποια άλλη χώρα να επενδύουν σε άλλη χώρα γιατί εκεί είναι πιο βολικά και είναι πιο αποδοτικό. Κάνουμε προσπάθεια όχι γιατί αυτός ο τομέας πλήττεται περισσότερο από το, από το οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε να διαφυλάξουμε στο μέγιστο βαθμό την παραγωγική διαδικασία. Θέλουμε να χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι θα πετύχουμε σωστή ισορροπία που είναι πολύ περίπλοκη. Δηλαδή, ανάγκη υποστήριξη παραγωγικών τομέων που είναι σημαντική, όπω των ελεκτικών μορφών ενέργεια, από τη μια και από την άλλη ανάγκη να υπάρχουν προστασίε, να... εκτεταμένε, που πρέπει να εφαρμόζονται σε ευρύτερε περιοχέ. Ε, και ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αν μίλησα λίγο περισσότερο από το χρόνο που είχατε διαθέσει. Ευχαριστώ. Όντως ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Τώρα ε, ε, είναι, ανοίγει ο γύρος της συζήτησης και θα σας έλεγα να καλύψουμε το θέμα αυτό μέχρι τις 10 και 10, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, αλλά οι ερωτήσεις αυτές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα δύο λεπτά σε διάρκεια. Ποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο, ο κύριος Σέρεν Άλτερ. Ίσως λοιπόν ε, ας ξεκινήσουμε ε, με ένα πολύ γενικό ερώτημα που αναφέρεται στην αποδοτικότητα των δαπανών διότι βλέπουμε ότι το 80% των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επανέρχονται στα κράτη-μέλη και πρέπει ε, να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα σε επίπεδο ενώσεως, σε επίπεδο κρατών μελών και αποδεκτών. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, εξετάζει κατά τομέα πολιτικής ε, τις επιδόσεις και τη διαχείριση των δαπανών και όσον αφορά την διοίκηση των ε, κρατών μελών η οποία εν μέρη χρηματοδοτείται από τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό ποια είναι η πορεία, ο κύριος Σέντεγκαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτησή μου αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε και ο τελευταίος ομιλητής. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πότε αυτή η διαδικασία της ε, εξετάσεως των ε, ε, επιπτώσεων της μαφίας μπορεί να οργανωθεί. Δηλαδή αναφέρομαι εις την κατάχρηση των κοινοτικών πόρων από τη μαφία και βλέπω ότι υπάρχουν ορισμένοι ο Νέστο Βιτορίτο, ο Χάνι Κάστρι, εκ των οποίων ο τελευταίος καταδικάστηκε για... Ε, ε για ε, εγκληματικές δραστηριότητες ε, ενώ είχε ήδη μία προηγούμενη καταδίκη δηλαδή πότε μπορεί κανείς να ελέγξει εάν έχει εμπλακεί κάποιος σε δραστηριότητες της μαφίας. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Ε, όταν εξετάζει κανείς ένα κύκλο ατόμων, καλό θα ήταν να ξέρουμε πόσα προ όσα τέτοια άτομα έχουν προκύψει όταν πρόκειται για μέλη της μαφίας άτομα τα οποία έχουν διαχειριστεί ε, κοινοτικούς πόρους υπάρχουν στατιστικές υπάρχουν ε, κατάλογοι και ε, ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς βεβαίως ο εισηγητής καταρχήν έχει το λόγο Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε και ε, αυτό που είπε ο κύριος Σλόιτερς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήταν πολύ σωστό. Αλλά εδώ μιλάμε για την... Ε, αποτελεσματικότητα και ε, πρέπει να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα ε, της χρήσεως του ε, ηλεκτρικού ρεύματος όπου είναι κάτι πολύ δαπανηρό. Βλέπουμε όμως εδώ ότι αναφερόμαστε και στην αποτελεσματικότητα για άλλους λόγους. Ανάφερε ο κύριος Σέντεγκαρντ αυτά που έχουν λεχθεί και στον τύπο, δηλαδή ε, τη διασπάθηση των δημοσίων πόρων ε, ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι ύψος ε, αριθμείται αυτή η διαφθορά σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και την αποτελεσματικότητα ενεργείας διότι εδώ μιλάμε για Ε, ε, πρόκειται για λεπτομέρειες μπορείτε να μου πείτε ακριβώς αν μπορούμε να αποκαλύψουμε την κατάσταση αν μπορούμε να επέμβουμε διότι ε, κάτι σε κάτι τέτοιο αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της Ιταλίας όσον αφορά τα δύο τελευταία πρωτόκολλα που είναι ένας τρόπος να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα ήταν ε, μπορείτε να μου πείτε ε, πώς ε, αξιολογείτε αυτόν τον τομέα. Μιλάμε για την αιωλική ενέργεια παραδείγματος χάρη. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ στον τομέα της αιωλικής ενέργειας όσο η Ιταλή εκπρόσωποι ε, είπαν ότι δεν χρησιμοποιείται τόσο η αιωλική ενέργεια. Αυτό οφείλεται στην εγκληματικότητα. Θα θέλαμε ε, συγκεκριμένες πληροφορίες. Ε, καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούν εντωμεταξύ να συνεννοηθούν οι εκπρόσωποι της Ιταλίας για το πώς πρόκειται να μιλήσει. Ε, όσον αφορά τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ε, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο οι Ιταλικές αρχές είναι αυτές οι οποίες πρέπει να ελέγξουν τα προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται και ε, πρέπει να μας αποδείξουν εάν έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για αποτελέσματα ελέγχου για τη χρήση των πόρων στην Νότιο Ιταλία. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πολύ υψηλό επίπεδο ε, παρατυπιών με τα ενεργειακά προγράμματα. Και εδώ αναφερόμαστε σε όλους τους τομείς ε, ενεργείας. Επίσης προσπάθησα να τονίσω κάτι που ελέγχθηκε από τον κύριο Στές δηλαδή ότι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από τα σχόλια της Λέγκα που συμμετέχει σε αυτή τη συνεδρίαση είναι ότι το πρόβλημα αναφέρεται ιδίως στην πράσινη ενέργεια και για διάφορους λόγους έχουμε λιγότερη συμμετοχή εις ε, την ε, ε, αιωλική ενέργεια τώρα από ό,τι στο παρελθόν και τουλάχιστον αυτό ισχύει για την Ιταλία. Μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας στην Ιταλία είναι λιγότερο εκτεθειμένοι εις την παράτυπη χρήση μετά το όλο ερώτημα του κυρίου Σόντεργαρτ. Θα πρότεινα η Ιταλική αντιπροσωπεία να εκφράσει την άποψή της επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παραγκόνε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν σεβαστήκαμε την διαδικασία Είχα πει στον κύριο ε, Στάση προηγουμένως ότι θα ήταν σκόπιμο να παρέμβουν και εκπρόσωποι της περιφέρειας. Ε, εγώ θα μπορούσα να δώσω, αν συμφωνεί ο Πρόεδρος, κάποιες απαντήσεις γενικού χαρακτήρα για το ρόλο που εμείς ε, παίζουμε και στη συνέχεια θα πρότεινα να δώσετε το λόγο σε όσους επί τόπου έχει εφαρμόσει όλα αυτά, δηλαδή στην περιφέρεια της Σικελίας, που έχει πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως ήδη αναφέρθηκε. Εγώ δεν νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους κινδύνους χρήσης των κοινοτικών πόρων Ε, των πόρων αυτών για την ελληνική ε, ε, ενέργεια. Η δίσδυση της μαφίας είναι γενικό πρόβλημα και αφορά όλους τους τομείς όλες τις περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να κερδίσει λεφτά. Το να σκεφτόμαστε ότι είναι μόνο η ολική ενέργεια θα ήταν μάλλον ανόητο. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό ε, μολύνει όλους τους παραγωγικούς τομείς και όλους τους επενδυτικούς τομείς. Από την οικονομία την ε, ε, ψηλή μέχρι το πιο απλό πράγμα. Τώρα, η δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι, να ενισχυθεί ακόμα, είναι το θέμα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ε, εφορία μας ε, για να μπορέσει να ερευνήσει καλύτερα το τι συμβαίνει, να καταστήλει την οικονομική εγκληματικότητα σε σχέση με τους ε, κοινοτικούς πόρους. Άρα και εκεί όπου αυτό συμβαίνει στον τομέα της αιωλικής ενέργειας. Τώρα όσον αφορά τις, ε, την αιωλική ενέργεια και την έλλειψη επενδύσεων ε, δεν σημαίνει αυτό πως η ενέργεια είναι, κινδυνεύει. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στο παρελθόν και άρα θα πρέπει να γίνει μια συστηματική μελέτη για να δούμε αν οι επενδύσεις που έχουν γίνει χρειάζεται να ε, ε, στηριχθούν για το μέλλον. Ε, τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες ερωτήσεις, θα είναι ίσως καλύτερο να παρέμβουν για τα συγκεκριμένα ερωτήματα εκπρόσωποι της περιφέρειας της Σικελίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλάτη, σας ευχαριστώ. Σύντομα και συνθετικά τα ενδιαφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας στον τομέα που εγώ παρακολουθώ στη Σικελία, όπως και σε όλους τους κερδοφόρους τομείς, δυστυχώς, και βέβαια η πράσινη οικονομία δεν είναι νέος τομέας. Φυσικά και ενδιαφέρεται το οργανωμένο έγκλημα για αυτά όλα. Όλους τους κερδοφόρους τομείς τους ενδιαφέρουν. Έχουμε δει περιπτώσεις, ε, δεν έχω βέβαια μαζί μου στατιστική μελέτη, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις και σχέσεις με τις νομαρχίες και το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν βγει στο φως ένα σωρό υποθέσεις και φυσικά εκεί αμέσως εκδώσαμε την ανάκληση της έγκρισης των εγκαταστάσεων και της χρηματοδότησης. Υπήρξαν επίσης ε, περιπτώσεις διαφθοράς αλλά που σε εμά η αλλαγή πορεία από την αιωλική ενέργεια στη φωτοβολταϊκή είναι μια αλλαγή πορεία που σχετίζεται με τη διαχείριση τη ε, περιφέρεια και βεβαίω οι αιωλικέ εγκαταστάσει είναι πολύ πιο κερδοφόρε από τι μικρέ και μέσε εγκαταστάσει φωτοβολταϊκή ενέργεια και είναι πολύ πιθανό εδώ να υπάρξει μικρότερο ενδιαφέρον από πλευρά του οργανωμένου εγκλήματο σε σχέση με τις ε, μεγάλες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν θέσαμε, εξάλλου υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που βγήκε στις εθνικέ και διεθνείς εφημερίδες, ήταν αυτός ο επιχειρηματίας που είχε επενδύσει στην ε, Αλκαμό 40-70 εκατομμύρια ευρώ στην ολική ενέργεια και εκεί το κράτος παρενέβη γρήγορα και η δικαιοσύνη και σήμερα αυτή η επιχείρηση που παράγει ενέργεια από αιωλική, από, την ολική ε, ενέργεια είναι στα δικαστήρια και από τα όσα έχουν προκύψει μέσα σε λίγους μήνες ε, έχει γίνει κατάσχεση του έργου και αυτή τη στιγμή τη διαχείριση έχει αναλάβει το Ιταλικό κράτος. Ε, συχνά Βεβαίω, το οργανωμένο έγκλημα εγκαθίσταται χρησιμοποιώντα τη διαφθορά και εμεί στην περιφέρειά μα, στη Σικελία προσπαθούμε να βάλουμε ε, ισχυρά όρια και να παρέμβουμε και σε το καθεστώς ε, αδειοδότησης. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα ευρωπαϊκά χρήματα, ενδιαφέρεται και για την αδειοδότηση, την πολοδομία, για την δημιουργία και την κατασκευή εγκαταστάσεων και εργοστασίων. Και εδώ παρενέβημε με ένα ισχυρό τρόπο. Ε, ξεκινήσαμε μια ολόκληρη σειρά ελεγκτικών δραστηριοτήτων επιτόπου, πράγμα το οποίο μας έδωσε ήδη αποτελέσματα και ελπίζω θα συνεχίσει να δίνει καρπούς. Δεν ξέρω αν ήμουν ε, πλήρη στην απάντηση που θέλατε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρίνο, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή όχι. Ε, ε, could you pay attention to Παρακαλώ, μπορείτε να ε, φροντίσετε τις ερωτήσεις του κύριου Σάντριγκάρντερ, ο οποίος ρώτησε τι συνέβη στον κόσμο εκεί. Ίσως μπορείτε να επαναλάβετε για να ε, απαντήσει ο κύριος Μαρίνο. Ναι, ίσως να υπήρξε πρόβλημα μετάφρασης. Να προσπαθήσω λοιπόν με τα φτωχά αγγλικά που είναι ίσως καλύτερα να τα πω στα αυτά παρά στα δανέζικα. Καταρχήν ρώτησα πότε εισήχθη ο κανονισμός ε, για την εξέταση των σχέσεων των ετούντων με τη μαφία γιατί έχουμε μια περίπτωση του Νοεμβρίου 2009 όπου συνελήφθησαν 15 άτομα, δύο εξ αυτών ε, καταδικάστηκαν και ενώ ένας από αυτούς το 2006 ήδη είχε καταδικαστεί για έγκλημα σε αυτόν τον ίδιο τομέα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το ερώτημα πότε εισήχθησαν αυτοί οι κανόνες για έλεγχο ε, σχέσεων με τη μαφία. Και έπειτα, αφού εισήχθη αυτός ο κανόνας, πόσες περιπτώσεις βρήκατε όπου υπάρχει σχέση με τη μαφία και για ποια πόσα μιλάμε. Κύριε Μαρίνο, μπορείτε να απαντήσετε. Ο κύριος Τζεράλντι. Λοιπόν, η υπόθεση αυτού του άρθρου στην εφημερίδα δεν τη γνωρίζω. Αυτό το άρθρο το γνωρίζω. Δεν ξέρω κανένα από τα δύο πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο, προσωπικά βέβαια. Δεν ξέρω πώς είναι πλάκι το άλλο άτομο στην όλη ιστορία. Ε, το ανέφερα, ανέφερα την υπόθεση αυτή στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Το 2009, όταν ανακαλύφθηκε ο δικαιός Νικάση μέσω της μαφίας έκαφη τεράστια επένδυση, παρενέβη, μεν, παρενέβη το κράτος και σήμερα αυτή η εταιρεία ε, διχειρίζεται το κράτος. Η σειρά των πρωτοκόλων και των μέτρων που δημιουργήσαμε σαν περιφέρεια της Σικελίας. Αυτά τα μέτρα λέγω αναφέρονται στο δεύτερο εξάμεινο του 2010 τα πιο σημαντικά μέτρα ελήφθησαν το δεύτερο εξάμεινο του 2010 και ισχύουν μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω, το θέμα Νικάστρη δεν συνδεόταν μόνο με, τα, με τους δημόσιους πόρους και τη χρήση αυτών αλλά με ένα σύστημα διαφθοράς για να πετύχει τις διάφορες άδειες. Γίνονται έρευνας και δεν είμαι πάνω σε αυτό το ιδεώδες άτομο να απαντήσω. Δεν αφορά μόνο τα δημόσια χρήματα ενδιαφέρον την Ικάρση, ήθελε, τον ενδιέφερε και να πάρει και τις άδειε. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, παρενέβημε την πρόσφατη περίοδο. Τα πρωτόκολλα μεγαλύτερη χρήση των μέσων κατά καταπολεμήσεως της διαφθοράς και της διείδησης της μαφίας σίγουρα ελήφθησαν το δεύτερο εξάμεινο του 2010 και μετά. Τις συγκεκριμένε υποθέσεις που ανακαλύψαμε αφορούν μικρές παρεμβάσεις στον τομέα της φωτοβολταϊκής ενέργειας 2000-2006 και της βιομάζας. για παρεμβάσεις περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και αμέσως βέβαια ήρθαμε σε επαφή με την Όλαφ και σταματήσαμε τις χρηματοδοτήσεις. Κινητοποιείται άμεσα ο μηχανισμός μέσω της, νομο, της νομαρχίας της ε, περιφέρειας, του νησιού. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση εδώ, παρόλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε να έχει συνεχιστεί, αλλά έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ότι ε, καλό είναι να παρουσιαστεί και η άποψη της ε, Europol και η διαθεσμική συνεργασία. Γι' αυτό και τώρα θα δώσω τον ε, λόγο στον κύριο Ότινγκ, εάν προέφερα καλά το όνομά του. Εξαιρετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε την Europol σε, αυτό το, σε αυτή την εκδήλωση και θα ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Europol και αναφερόμαστε εις ε, τις ε, φορολογικές απώλειες ε, και δεν είμαστε σε θέση να ερευνήσουμε την κατάχρηση πόρων. Αυτό γίνεται από την Εθνική Αστυνομία αλλά συμβάλλουμε εις την αστυνομική συνεργασία για την εφαρμογή του νόμου. Η Europol λοιπόν είναι είναι ε, ε, ε ε, το ε, ε, σκέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που αναλαμβάνει την εφαρμογή του νόμου και καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα νέα έδρα στην Ολλανδία και έχουμε πάρα πολλούς ειδικού οι οποίοι συντονίζουν τους εμπειρογνώμονες σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε χώρες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην Κολομβία, στην Αμερική, στην Ισλανδία. Υπάρχει μία συνεργασία διαφόρων αρχών τελωνιακών, αστυνομικών σε ένα ευρύ πλαίσιο. Ε, εξετάζουμε περίπου 13.000 περιπτώσεις ετησίως, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ επιτυχείς στην, ε, στο συντονισμό της συνεργασίας και ε, ε, ε, η Europol συντώνησε παραδείγματος χάλιν και την, τις προσπάθειες της Νορβηγίας μετά το γεγονός εφέτος, τον, εφέτος το καλοκαίρι όπου σκοτώθηκαν 69 άτομα Επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι έχουμε όλα τα στοιχεία μας σε αναλυτικούς φακέλους δεδομένων. Ένα εξ αυτών ονομάζεται SMOC γιατί αναφέρεται σε την φοροδιαφυγή στο τομέα του καπνίσματος και έχουμε και ένα φάκελο σχετικά με την ε, φοροδιαφυγή για το ΦΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πέραν αυτών και ε, μία ε, πολύ πιο περίπλοκη φοροδιαφυγή για το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν της Ιταλίας ε, οργανώνεται από πολλές εγκληματικές ομάδες συμμορίες οι οποίες προσπαθούν να ε, συγκαλύψουν τα κέρδη των συμμετεχόντων στα, ε, ε, σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες διότι παρουσιάζουν καταρτίζουν μια εταιρεία η οποία χρωστάει ΦΠΑ και μετά διαλύεται και μένουν τα χρήματα στην τσέπη τους και δημιουργείται μια άλλη εταιρεία. Αυτό όμως είναι μόνο ένα εκ των προβλημάτων σε ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό περιπτώσεων και γι' αυτό μπορώ να σας πω το εξής για την τωρινή περίοδο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεταξύ των εγκληματιών μία διεθνή συνεργασία που τους επιτρέπουν να αναπτύσσονται ε, ε, διεθνώς σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ χωρών ε, και οι συμμορίες αυτές δεν αντιμάχονται μία την άλλη αλλά συνεργάζονται. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός αλλά έχουν ε, ε, συμμετοχή και στους πόρους και στα κέρδη. Ε, γι' αυτό και οι αστυνομικές ε, αρχές πρέπει να συντονίζονται, να διδάσκονται από τα λάθη μία της άλλης και επίσης οι, ο, οι εγκληματικές ομάδες επενδύουν στις δραστηριότητες παρεμφερών οργανώσεων και βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ε, ε, εγκαταστάσεις σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους και υπάρχει μία διαδικασία CP42.000 όπου βλέπουμε ότι διάφορες οργανώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητες και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και σε λιμάνια όπως η, ε, το Αμβούργο και το Ρότερνταμ και ε, ειδικεύονται σε τομείς όπως ο ΦΠΑ. Υπάρχει εδώ ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα διότι υπάρχει συνεχής προσαρμογή μπορείτε ας πούμε να ασχοληθούν τη μία μέρα με ε, το ΦΠΑ ε, για την εμπορία των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. την επόμενη μέρα με τις ε, κινητές ε, συσκευές τηλεφωνίας είναι πάρα πολύ δραστήριε και πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί εάν δεν καλύπτεται από τα κράτη-μέλη και υπάρχουν κενά διότι μόλις υπάρχει ένα κενό οι εγκληματικές αυτές αυτές οργανώσεις εποφελούνται. Υπάρχουν δέκοι κοινοτικοί πορεί οι οποίοι χρηματοδοτούν την ε, ε, οργάνωση ε, χρηματοδοτούν τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ΙΣΕΚΑ από την DG Home και ε, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ISEC ε, ε, είναι της αρμοδιότητος της Europol και βλέπουμε ότι είχαμε δημιουργήσει ένα σύστημα καταπολεμήσεως των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Βλέπουμε όμως ότι τώρα το σύστημα έχει αλλάξει και έχουμε αποκλειστεί από χρηματοδότηση και το πρόγραμμα ISEC ε, ε, θα πρέπει να ε, μπορέσει να συντονιστεί με την ε, ε, με την Europol ε, γιατί δεν θα πρέπει να αντιμάχεται τα συμφέροντα της Europol. Ένα σύνολο κρατών με επικεφαλή στη Ρουμανία χρηματοδοτήθηκε με ένα πρόγραμμα με βάση το Βουκουρέστι στο οποίο έπρεπε να συμμετάσχει και η ε, Europol που είναι η υπεύθυνη για ε, την ε, αστυνομική συνεργασία. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει τώρα μία νέα οργάνωση η οποία επικαλύπτει τις δραστηριότητες μας με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να προστατεύουμε προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από εγκληματικέ ενεργησής και ε, γι' αυτό είχαμε ε, ε, είχαμε συμμετάσχει στην, στα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της πλαστο, των πλαστών ευρώ και ε, εκεί πάλι ο συντονισμός δεν ήταν τόσο ε, ικανοποιητικός. Ε, τέλος υπάρχει ένα πρόγραμμα της Γενικής Διευθύνσεως επιχειρήσεων όπου βλέπουμε ότι οι αστυνομικές αρχές δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας και υπάρχει μία διασπάθηση ε, και σπατάλη των χρημάτων ε, διότι δεν μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τα προγράμματα ε, και πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Ποιες είναι λοιπόν οι συστάσεις μας για να μην κατακρίνουμε μόνο. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να καταρτιστεί ένα ταμείο για την προώθηση της εσωτερικής ασφαλείας κατά τρόπον ώστε να μπορέσει αυτή να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να χρησιμοποιηθούν ευέλικτοι οργανισμοί χρηματοδοτήσεων ε, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις αρχές. Επίσης θα πρέπει η Europol να συμμετέχει στην διαχείριση των πόρων αυτών και να συμβάλλει πιο επικοδομητικά στην διαχείριση των ε, ευρωπαϊκών πόρων. Ε, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το οποίο θα συνεργάζεται με την Ευρωπόλ και ε, θα καταρτίζει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων των δράσεων διότι ε, η Ευρωπόλ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει ε, θα πρέπει να μπορέσουν να έρχονται στις ε, ε, συναντήσεις να μπορέσουν να συντονίζουν τις ενέργειες διότι αν κράτη-μέλη δεν έχουν πόρους για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις αυτές θα μπορούσε η Ευρωπόλ να βοηθήσει αλλά τώρα η χρηματοδότησή μας στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένη. Πού καταλήγουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι σχετικά με ε, την ε, ε, ε, ε, το θέμα της φοροδιαφυγής ή στο ΦΠΑ προχωρούμε ικανοποιητικά και σε πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι η αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ δεν είναι φοροδιαφυγή και κακή χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει όμως να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας τα, ε, τις υπάρχουσες δυνατότητες και τις δυνατότητες της Ευρωπόλ. Και η Europol γι' αυτό θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαχείριση αυτών των πόρων για να μην υποθάλπονται οι ενέργειες της και να συμμετέχει περισσότερο εις ε, τους, ε, ε των ευρωπαϊκών πόρων ε, για να μπορέσει να επανέλθει στη θέση την οποία είχε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα επανέλθουμε λοιπόν σε όλα αυτά που μας είπατε. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Αντώνιο Περγκολέτσι από την ΜΚΕΟ. Λέγκα Αμπιέντε, Παρατηρητήριο για την νομιμότητα και το περιβάλλον. Έχετε το λόγο. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας ε, για σήμερα. Πρόεδρε, σε εσά ευχαριστώ και σε όλους όσους οργάνωσαν αυτήν εδώ την πρωτοβουλία. Όπως ξέρετε εγώ συμμετέχω σε ένα ΜΚΟ που μελετά τη διάφορα θέματα ε, σε σχέση με την νομιμότητα και την ε, εγκληματικότητα. Προσπαθούμε δηλαδή να ε, μπορέσουμε να σταματήσουμε κάθε παράνομο φαινόμενο το οποίο έχει σχέση με το περιβάλλον να πω ότι η ολική ενέργεια ε, μαζί με τα άλλε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι το μέλλον τη Ιταλία και τη Ευρώπη των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα από του λίγου τομεί που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη. Ε, μιλάμε για τεχνολογική ανάπτυξη και κυρίω την απεξάρτηση από, τις, από τα στέρεα καύσιμα. Ε, Όλα αυτά βεβαίως ε, μπορεί να παρεμποδίσουν και να διακόψουν ε, ε, ιστορικά συμφέροντα, πράγματα τα οποία μπορεί να οδηγήσει σε παρέμβαση. Γι' αυτό και υπάρχει η διείσδυση της εγκληματικότητας στις νέες πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχει και το κράτος. Υπάρχει το κράτος και εμείς μαζί η ΜΚΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβουμε ώστε αυτά τα φαινόμενα να μπορούμε να τα σταματήσουμε θα πρέπει λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε ε, καλά, αλλά ε, να μην καταλήξουμε στα λάθος χέρια. Στην αναλυτική μας δραστηριότητα απέναντι στα εγκληματικά φαινόμενα, ήδη από το 2007 έχουμε ασχοληθεί και αποδείξαμε το ενδιαφέρον των διαφόρων ε, συμμοριών της μαφίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για την υδροελεκτρική ενέργεια αρχικά. Εκεί ας πούμε το ενδιαφέρον στην Καλαβρία των ε, μαφιόζων για την αιωλική ενέργεια και την υδροελεκτρική έχει εκδηλωθεί από το 2007. Αλλά παρενέβησαν και οι δυνάμεις της τάξης εισαγγελία. Γίνονται δηλαδή συγκεκριμένες ε, ανακρίσεις και έρευνες. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είναι γεγονός. Στην Ιταλία το ξέρουμε πάρα πολύ καλή, είναι μια χώρα της μαφίας. Είναι μια χώρα όπου ορισμένε περιοχές, κυρίως στην, στην Νότια Ιταλία, ελέγχονται από την μαφία συνολικά και γενικά. Έχουμε ήδη φτάσει σε, έχουν φτάσει σε θέσεις πάρα πολύ ισχυρέ, έχουν συγκεντρώσει χρήματα και έχουν προβληθεί σε ένα σενάριο εθνικό και διεθνές τα άτομα για τα οποία μιλούσαμε προηγουμένως είχαν ε ε, ε, ε, μαφιόζικες δραστηριότητες στο Βέλγιο, στη Μάλτα και σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες. Δεν μιλάμε για μια μαφία όπως την έχουν παρουσιάσει παλιά η τηλεόραση, ότι δηλαδή είναι ένα φολκλωρικό φαινόμενο. Είναι ένα χαρακτηριστικό οικονομικό φαινόμενο που λειτουργεί σε διεθνή, σε διεθνή κλίμακα αυτή τη στιγμή. Οι διάφορες μαφίες είναι μόνο όμως ένας κρίκος της αλυσίδας. Είναι μια περίπλοκη αλυσίδα όπου συμμετέχουν ε, προσωπικότητες ε, με διαφορετικό εγκληματικό κύρος ε, επιχειρηματίες, ε, δημόσιοι υπάλληλοι, ε, πολιτικοί. Δυστυχώς το φαινόμενο της διαφθοράς, της σύνδεσης δηλαδή μεταξύ της, της οργανωμένης εγκληματικότητας και της δημόσιας διοίκησης είναι ακριβώς ο, ο, ο πυρήνας του θέματος. Πρέπει δηλαδή να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες και εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που μετά δίνουν το πράσινο φως σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι από την άποψη του modus operandi το οργανωμένο έγκλημα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας δεν κινείται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους τομείς. Η ιστορία ελέγχουν την περιοχή ε, παρεμβαίνουν ε, στις, στους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς, ε, λειτουργούν στους διάφορους οικονομικούς τομείς, προσπαθούν να επηρεάσουν την αγορά εργασίας και να ρυθμίσουν κάθε πτυχή της. Ακριβώς θέλουν να διώξουν την υγιή οικονομία, να καπελώσουν έναν τομέα και να φτιάξουν μετά παρασιτικές δραστηριότητες που θα τους φέρουν κεφάλαια και τα οποία θα επενδύσουν σε διάφορες δραστηριότητες και νόμιμου τύπου. Συχνά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να δει πού πήγαν τα χρήματα, τις ροές, τις οικονομικές. Και εκεί θα πρέπει κανείς να παρακολουθήσει τη ροή των χρημάτων, όπως έλεγε και ένας σπουδαίος εισαγγελέα, ο οποίος ε, ε, δολοφονήθηκε από τη μαφία, ο Τζοβάνι Φαλκόνε θα έπρεπε δηλαδή να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, να παρακολουθήσει τα χρήματα, πώς κινούνται, πώς καταφέρνουν δηλαδή να επιβληθούν στην περιφέρεια και μετά να επεκταθούν και πιο πέρα. Ο Ρομπέρτο Καρπινάτο που είναι εισαγγελέα και που είναι και ένας από τους συζητητές θα μπορέσει να σας το εξηγήσει και καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά τα εγκληματικά συστήματα και πώς δρούν και κυρίως πώς καταφέρνουν να επηρεάσουν τις ε, διοικητικές επιλογές. Το, essere... Ε, και από την άλλη πλευρά θα μπορούσε, δεν, θα, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά γιατί πρόκειται για λογικά άτομα όπως έλεγε ο Φαλκόνη και προσπαθούν να καρποθούν κάθε πηγή δημόσιας χρηματοδότησης. Στον τομέα αυτών είναι τριών ειδών οι χρηματοδοτήσεις, δηλαδή κεφάλαια, συμφέροντα και μέσω των πράσινων προσπιστοποιητικών συμφέροντα. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ροές των δημοσίων επενδύσεων, των δημόσιων χρηματοδότησης προς συγκεκριμένους ε, λογαριασμούς. Μόνο, από το, μόνο το 2006, αν δεν έκανα τα λάθος στους λογαριασμούς, πάνω από 225 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάει σε τέτοιους είδους δραστηριότητες ε, με βάση τον νόμο για το περιβάλλον. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να μπορούμε να πούμε πόσα δημόσια χρήματα κατέληξαν στα ταμεία του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν αποφάσεις πρωτοβάθμιες, αποφάσεις που έχουν συνδυάσει και ποινές που φτάνουν σε εκατοντάδες ε, χρόνια κάθριξης. Υπάρχει δηλαδή η δικαιοσύνη και η λειτουργία, αλλά μιλάμε για πρωτοβάθμιες αποφάσεις. Έχουμε άλλους δύο ε, βαθμίδες δικαιοδοσίας και πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα υποκείμενα και ποιες είναι οι ευθύνες του κάθε φορά. Φυσικά ε, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετράμε τη νέα στρατηγική των μαφιών, δηλαδή να μπαίνουν σε πολύ ψηλής τεχνολογίας τομείς. Συνήθως ε, ασχολούνταν με διάφορους τομείς ε, που δεν χρειαζόταν μεγάλη τεχνολογία, δηλαδή τρόφιμα και τσιμέντο. Και έχουν κάνει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της χώρας μας. Αν δείτε ας πούμε τα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν στην επικράτειά μας και στις στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες οικονομικές αυτοκρατορίες που έχουν ε, στην ουσία κάνει συμβάσεις με το διάβολο, έχουν κάνει συμφωνίες με το διάβολο για να μπορέσουν να κατασκευάσουν αυτά τα έργα. Δεν είναι πρόβλημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ολικής ενέργειας, αλλά είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα το οποίο απλώνει τα πλοκάμια του παντού. Τα κίνητρα για να μπορεί κανείς να μπει σε αυτό το τομέα ήταν ε, πάρα πολλά. Ε, Καταρχήν δεν υπήρχε δυνατότητα προγραμματισμού της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπήρξε μέχρι πέρσι το 2010 μια πραγματική στρατηγική εθνικού επίπεδου που κατά κάποιο τρόπο να συνοδεύει την ανάπτυξη της ολικής ενέργειας. Όλα έγιναν πέρα από οποιοδήποτε εθνική, εθνικό κανόνα, οπότε στην ουσία γίνανε όλα χαοτικά. Δεν έφτασαν εγκαίρως ε, και μέσα ελέγχου για αυτό το τομέα, αλλά σιγά σιγά η δυνατότητες καταστολής αυτού του φαινομένου εκδηλώνονται και εμφανίζονται. Όπως σας είπα, οι συμμορίες της μαφίας έχουν τεράστια κεφάλαια να χρησιμοποιήσουν και να επενδύσουν και καταφέρνουν να ρυθμίσουν, όπως έλεγα και προηγουμένως, τα μέσα της αδειοδότησης μέσω της διαφθοράς, ε, που είναι το πραγματικό πρόβλημα. Σε μια από τις τελευταίες έρευνες όπου έχουμε αποτελέσματα, αυτό που αφορά την Πούλια, την ε, έρευνα Ventus για την περιοχή της Πούλια, όπου επρόκειτο για τη δημιουργία ενός αιωλικού πάρκου μέσα στο πάρκο της ε, ε, αλτα ΜΟΥΡΤΣΙΑ, δηλαδή στην ουσία δεν είναι μόνο φαινόμενο απορρόφησης χρημάτων ε, αλλά και περιφερειακά θέματα από άποψη οικονομική γιατί αυτό έγινε μέσα σε ένα πάρκο φυσικό, υποτίθεται προστατευόμενο. Θα θυμάστε τον περασμένο Ιανουάριο την Μεσίνα, την υπόθεση της Μεσίνας που οδήγησε και σε κατάσχεση 25 εκατομμυρίων ευρώ, δεν αναφέρω νόματα γιατί ακόμα τρέχει η ε, διαδικασία Πάντως ε, πρόκειται για σύνδεση με τον Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, που έναν άνθρωπο με τον οποίο, για τον, ο συνδεόταν με εκείνα τα οποία ε, αναφέρθηκαν προηγουμένως. το πρόσωπο του εργολάβου, που είναι το σημαντικό πρόσωπο, γιατί είναι αυτός που, αν και δεν έχει ε, γη, όπου να φτιάξει δηλαδή τις αιωλικές... Ε, το, το υλικό πάρκο, αν και δεν είχε χρήματα, κινείται μέσα σε μια επικράτεια μέχρι ότου να πάρει όλες τις άδειες. Άπαξ και πάρει όλες τις άδειες και τη δέσμευση της, για τη χρήση της γης, από τη στιγμή που έχει το πακέτο το πουλάει σε μια πολυεθνική σε κάποιον άλλον ε, επιχείρηση. Όχι απαραίτητο πολυεθνική. Αυτή η ελευθερία δράσης του εργολάβου, ας πούμε, του αυτού που, που είναι υπεύθυνο για το έργο και είδαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει ανοίξει παραθυράκια για ένα μεγάλο φαινόμενο αδιαφάνειας και η επέκταση αυτών των ατόμων που δεν έχουν κεφάλαια και που πουλάνε ένα τελειωμένο πακέτο σε άλλες επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να σταματήσει μέσω ας πούμε των ε, λογαριασμών τους, των τραπεζικών ή εν πάση περιπτώσει μέσω της ελευθερίας δράσης αυτών των ανθρώπων που συχνά είναι ε, ε, επιχειρηματίες, επιχειρηματίες που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, θα χρειαστεί να διαχειριστούμε επενδύσεις για 10 δις ευρώ. 10 δις ευρώ τα οποία έχουν προορισμό την ανανεώσιμη ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πάρα πολύ. Να δώσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα. Καλαβρία. Για να σας δείξω το πρόβλημα της διείσδυσης ε, του οργανωμένου εγκλήματος σε μια περιφέρεια όπως αυτή της Καλαβρίας. Σε 18 ε, αιωλικά πάρκα, σε όλα γίνεται έρευνα εισαγγελική. Εκεί όπου άμεσα υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου άμεσα συμμετέχουν οι συμμορίες της, της μαφίας ή άτομα που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται με τις συμμορίες. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι η γεωλική ενέργεια ή οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά είναι η μαφία και οι μαφίε που θα πρέπει να τι σταματήσουμε. Και μάλιστα αυτό με μεγάλη ισχύ. Η αιωλική ενέργεια είναι ένα από τα διάφορα που μπαίνουν στο καλάθι του οργανωμένου εγκλήματος και δεν είναι το μεγαλύτερο. Παρ' όλα αυτά ε, χρειάζεται να γίνει μια ε, ανάγνωση ίσως και υπερβολική. Προσπαθούμε να δώσουμε και να ποσοστοποιήσουμε το φαινόμενο από την άποψη των, ε, την οικονομική. Και έχουμε συνδυάσει, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας, την Ιταλία, τις έρευνες που αφορούν ε, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις, ε, τις αγγελικές έρευνες για το τσιμέντο, τα ζώα και τη νεολική ενέργεια. Και μιλάμε για 5,9% διαλική ενέργεια από όλα αυτά. 5,9% είναι οι εισαγγελικέ έρευνε που αφορούν όχι απαραίτητο στη συμμετοχή των συμμοριών, αλλά απάτε ε, διαφθορά και ούτω καθεξής. Ενώ για το τσιμέντο έχουμε μόνο τις περιπτώσεις όπου είναι βεβαιωμένη η συμμετοχή της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. 5,9 λοιπόν είναι η ολική ενέργεια σε αυτές τις αγγελικές έρευνες για να δείτε ποιο ε, είναι το μέγεθος του οργανωμένου εγκλήματος εδώ στην να κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια οικονομική δυνατότητα τεράστια. Συνδέονται όλα αυτά με τη μαφία και θα πρέπει να, προσπαθούν να καθορίσουν τις μικρές ε, τοπικές πραγματικότητες. Καταρχήν τον δημόσιο τομέα τον ε, μικρό τοπικό παράγοντα. Βάζουν τα λεφτά φτάνουν τα δημόσια λεφτά σε ένα μικρό μέρος που έχουν τη δυνατότητα να διαφθείρουν ολόκληρο το σύστημα, να δημιουργήσουν αδιαφάνεια και σίγουρα και πολύ συχνά αυτά τα δημόσια χρήματα τα οποία ε, στέλνονται ξαφνικά σε μια μικρή περιοχή όπου η ε, παρουσία ενός τοπικού παράγοντα και του του πελατειακού του δικτύου μπορεί να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού και μπορεί όντως τα δημόσια χρήματα που στόχο έχουν την ανανεώσιμη ενέργεια να καταλήξουν στα λάθος ε, χέρια. Χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Μιλήσατε πριν για πρωτόκολλα συνεννόησης. Αυτό σημαίνει πως και οι διάφορες κατηγορίες που είναι θύματα θύματα αυτών των φαινομένων, ε, όπως οι, οι, υγιείς ε, επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο τομέα και που είναι θύματα αυτής της οργανωμένης εγκληματικότητας. Ε, ο Πρόεδρος διακόπτη. μπορείτε να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ. Φινίρε, Σιλβουπλέ. Ναι, να κλείσω λέγοντας ότι χρειάζονται περισσότερη έλεγχη, περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στις ε, Ιταλικές αρχές και τις Ευρωπαϊκές, ώστε να μην πληγεί ένας τομέας ο οποίος αντίθετα χρειάζεται να στηριχθεί. Το γεγονός ότι βλέπουμε και από τις διαφάνειες μια κάθετη αύξηση της ε, παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από τις επικράτειες στη Νότια Ιταλία ε, δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό, είναι η θετική κατεύθυνση. Αυτή θέλουμε από εδώ, είναι κόντρα στην ε, θέρμανση του πλανήτη κτλ. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε και να προσέξουμε ώστε τα χρήματα να μην καταλήγουν στα λάθο χέρια. Το πρόβλημα είναι η μαφία πρέπει να μπορέσουμε να παρέμβουμε ε, αποτελεσματικά για να τη σταματήσουμε γιατί λειτουργούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε όλους τους άλλους τομείς. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω όλε αυτέ τι προσπάθειες ε, να συμβάλλουν στο να αποφεύγουμε να φτάνουν σε λάθο χέρια τα λεφτά. Θα ήθελα να αφιερώσουμε 15 λεπτά λίγο πολύ προς συζήτηση, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και την απαλλαγή του Συμβουλίου. Ο κ. Σίτταλα, η κυρία Κρέσλε, ο εισηγητή βέβαια στο τέλος. Ορίστε. Κ. Μπαλσίτης. Έχουμε όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Οπότε κλείνουμε τον κατάλογο. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας. Ο κ. Ιταλά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους προλαλήσαντες για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή διότι πρόκειται για ε, πολλές πληροφορίες οι οποίες είναι συνταρακτικές ε, Σχετικά με την Ευρωπόλ έχω δύο ερωτήσεις. Πρόκειται για συγκεκριμένα ποσά. Ο, σχετικά με την όλα αυτό ο, την Europol και το Κοινοβούλιο πώς μπορούμε ε, από κοινού να προβλέψουμε μία στενή συνεργασία και να καταπολεμήσουμε την, ε, ε, το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης η Ευρωπόλ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ερευνές ή έχει απλώς ένα συντονιστικό ρόλο. Ε, η κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ να μας δώσετε το χειρόγραφό σας διότι δεν το έχω στα έγγραφα είπατε ότι ε, εάν υπάρχει διασυνοριακή ε, φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία. Πρώτη φορά ακούω ότι δεν υπάρχει γιατί νόμισα ότι χρηματο... χρησιμοποιώντουσαν τα στοιχεία που υπάρχουν εις ε, τις τράπεζες δεδομένων διασυνοριακά και ε, σχετικά με τη Γερμανία έχουμε τώρα στη Φραγκφούρτη μία πολύ σοβαρή περίπτωση για τα δικαιώματα που καταβάλλονται για την εμπορία ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και την παρακολουθούμε. Επίσης υπάρχει συνεργασία με μία υποργάνωσή σας, τη ΣΕΠΟΛ και ζητήσαμε να συνεργάζονται οι Ευρωπόλ με τη ΣΕΠΟΛ. Τι γίνεται με αυτή τη συνεργασία, ο κύριος Βαρίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το θέμα το οποίο συζητούμε. Ε, δεν είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθούμε γιατί εγώ νόμιζα ότι ήμουν ε, σε ε, μία επιτροπή ήτρε διότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων ήταν πολύ ικανοποιητικά. Το ερώτημα όμως είναι πόσα από τα 300 εκατομμύρια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί παράτυπα, παράνομα και κοιτάζω προς τα πίσω παρόλο που άκουσα ότι πρόκειται να επενδυθούν επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας στα, εντός των επομένων ετών και βεβαίως η, το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι ε, περίεργο ότι θα ασχοληθεί με τον τομέα αυτό. Όχι μόνο για τα χρήματα αλλά και για επέμβαση στην πολιτική ζωή των χωρών και εδώ δεν αναφέρομαι ειδικό στην Ιταλία. Υπάρχουν παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε πάντοτε τι ακριβώς συνέβη και αυτό με κάνει να σκέφτομαι όλα αυτά τα θέματα τα οποία εκκρεμούν και τα οποία και η Επιτροπή αυτή και η Όλαφ και η ε, Europol θα έπρεπε να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι όντως θα χρησιμοποιηθούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Τώρα δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από το ελεγκτικό συνέδριο για τον αριθμό των περιπτώσεων όπου έχουν ξεκινήσει οι έρευνες στο χώρο αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της ακρόασης διότι το πρόγραμμα δεν, είναι, δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και να καταρτήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να διευκολύνει τη ζωή των καλών ανθρώπων και εδώ και στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τελικά στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω τις ερωτήσεις αλλά να θέσω και ένα ερώτημα προς δύο διαφορετικούς. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Φαζάκας. Ακούσατε τα όσα υπόθηκαν τι σχεδιάζει να κάνει το ελεκτικό συνέδριο. Θα συντάξετε μια ειδική έκθεση για τον τομέα. Θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα. Φαίνεται ότι το ζήτημα είναι σοβαρό. Και θα εκτιμούσαμε βέβαια τη βοήθεια του ελεκτικού συνεδρίου. Κάνατε μια, μια πολύ ωραία γενική εισαγωγή καλή τροφή για τη συζήτηση, αλλά θα μπορούσατε πιο συγκεκριμένο σχετικά με τις δραστηριότητε που θα εφαρμόσετε. Μετά, κύριε Σλάουτερς, παρόμοια ερώτηση. Εξεπλάγιν που σας άκουσα να δίνετε απάντηση στο ερώτημά μου του πρώτου γύρου. Είπατε ότι μιλάμε για 300 εκατομμύρια, διενεργούνται έρευνες, κυρίως είναι ευθύνη των κρατών μελών αυτή, ναι, σωστό, μιλάμε για κοινή διαχείριση και την τελευταία δεκαετία σε όλες τις διαδικασίες απαλλαγής είπαμε ότι η κοινή διαχείριση αποτελεί πρόβλημα. Πινκ-πονγκ μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Εμεί σαν Επιτροπή Ενέχου Προπολογισμού πάντα προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα επομίζονται τι ευθύνε του. Ότι θα πρέπει να επομιστούν τι ευθύνε του και να προσπαθήσουν να λάβουν εγγυήσει από τα αρμόδια Υπουργεία ότι διενεργούν έρευνε. Ακούσαμε από τι εκπροσώπου κελίας ότι αναλήφθησαν κάποιε πρωτοβουλίε, τα δύο πρωτόκολλα, παραδείγματο χάρη. Χαίρομαι που έγινε αυτό και θα ήθελα να σα ρωτήσω εάν υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε. Αν τι έχετε, παρακαλώ στείλτε μα σχετικά έγγραφα. Θέλουμε γραπτέ πληροφορίε. Θα μα ωφελούσαν. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέποντας την κατάσταση ε, τίποτα θεωρείτε ότι δεν πάει πολύ στραβά. Ακούγοντας αυτά που υπόθηκαν, τι θα, κάνουν τι θα κάνει η Γενική σας Διεύθυνση. Σε εσύ τι συμπαράσματα θα καταλήξει από τις πληροφορίες αυτές που ακούσαμε. Τι θα πείτε ότι επισήμως δεν γνωρίζουμε τίποτα για όλα αυτά. Δεν ξέρουμε που πάνε τα χρήματα. Πού είναι η δική σας ευθύνη, ποια ευθύνη θα επομιστείτε, όχι προσωπικά, όταν λέω εσείς, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τον κύριο Έρτινγκ και μετά θα δώσω το λόγο και στον κύριο Φαζάκας και μετά στον κύριο Σλόιτερς. Και μετά ο κύριο Μπουργολής, αν θέλει να απαντήσει, θα του δώσουμε το χρόνο. Ο κύριο Όλτινγκ είναι ο πρώτος. Θα είμαι σύντομος, προς να είμαι σύντομος. Προς το φιλανδικό ερώτημα να απαντήσω δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό. Πρέπει να ακολουθήσουμε στατηγική που χρειάζεται διάφορους φορείς. Αναφέρατε το ελεκτικό συνέδριο, την Όλαφ και την Ευρωπόλ, που θα μπορούσαν να καλά παραδείγματα για ένα ξεκίνημα. Είναι πολύ καλή δυνατότητα για μας να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Ρωτήσατε αν θα έπρεπε να έχουμε εξουσία για έρευνες. Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε στα κράτη-μέλη πραγματικά θέλει κάτι τέτοιο, άρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε καλοί να στο συνεντονίζουμε και μπορούμε να πετύχουν πολλά έτσι. Ο μόνο τομέα όπου πιστεύω ότι ίσω να μην. ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον δυνατότητα να κάνουν περισσότερα θα ήταν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να βλέπουμε τον οθόνη του υπολογιστή και να μην μπορούμε να κάνουμε κάποιο εικονικό έλεγχο στον κυβερνοχώρο. Χρειάζεται μια προσαρμογή εκεί αλλά πραγματικές ερευνητικέ εξουσίες δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτή τη φάση. Για το γερμανικό ερώτημα βέβαια μπορεί να έχετε ένα αντίγραφο του, ένα αντίγραφο του εγγράφου. Δεν μπορεί το ΣΕΡΚΑΣ να ενταχθεί στην Ευρωπόλ διότι υπάρχουν πολλέ ε, χώρες ε, υποψήφιε και η Τουρκία είναι επίσης εταίρο. Δεν θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι το εφεύραμε με έναν τρόπο που κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνει και η Ευρωπόλ. Και πάνω από 95% των κρατών μελών στο κέντρο αυτό θα γίνουν κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκτός από την Τουρκία φαντάζομαι. Στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Αύριο θα συναντηθώ με τους Αμερικανούς και την DG Home και ελπίζω ότι μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό. Γιατί είναι ανόητο. Μετά, εάν υπήρχε δυνατότητα όσον αφορά τις απάτες να είναι πιο καλά προσαρμοσμένο, να προσαρμόσουμε το σύστημα. Είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες. Αυτή είναι και η δική μου εμπειρία. Έχουμε 27 χώρες. Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 15. Αλλά ο ίδιος είναι και στο διαπράτη το αδίκημα και αν δεν συνεννούμαστε με τις χώρες δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες και τα τεράστια έσοδά τους που πάνε στο Ντουμπάι, στο Πακιστάν και αλλού. Πάρα πολύ γρήγορα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν συζητήσουμε τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ να υπάρχει υποχρεωτική κοινοποίηση από τα κράτη-μέλη σε κάποιες υποθέσεις που έχουν προτεραιότητα διότι τώρα είναι στη διακριτική του ευχέρεια να το κάνουν. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κάτι Δεν έχουμε κίνητα να του υποχρεώσουμε. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Για να βοηθήσουμε όμω χρειαζόμαστε τι πρώτε ύλε. Αυτά έχω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φαζάκα, κύριε Φαζάκα, μπορείτε να μα πείτε ποια είναι η αρχική σα ε, εντύπωση. Τι μπορεί να κάνει το ελεκτικό συνέδριο μετά από αυτά που ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεργαζόμασταν πάντα. Και γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος Συνοψίζω. Μήνυμα ελήφθη. Αλλά ας πω περισσότερα. Καταρχάς ευχαριστώ που εκτιμήσατε δεόντως την παρουσίασή μου. Όπως είπα στην αρχή, έχοντας λάβει την πρόσκλησή σας, σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε καλύτερα στη συζήτηση. Και μετά είπαμε το καλύτερο θα ήταν να σας δώσουμε επισκόπηση των δραστηριοτήτων μας. Και ιδιαίτερα το πώς όχι μόνο να διαφυλάσσουμε την νομιμότητα και τον τακτικό χαρακτήρα, αλλά την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν είναι ερευνητικό φορέα, ούτε διοκτικό φορέα. Κάνουμε του ελέγχου μα σύμφωνα με τα σχέδιά μα. Και είσαστε βασικοί εμπλεκόμενοι εσεί. Και κατόπιν αιτήματό σα πάντα ήμασταν ανοιχτοί. Θέλαμε να ακούμε τα αιτήματά σα. Όσον αφορά την Ιταλία, βλέποντας τι έχουμε κάνει και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, δεν έχει έλεγχος επίδοσης όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου αλληλεγγύης στην περιοχή Αμπρούτσιου. Εγώ είμαι εισηγητής για έκθεση. Απόδοση αποτελεσματικότητα των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας έχει δρομολογηθεί έκθεση. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το στόχο και το θέμα ή να αρχίσουμε καινούργια έκθεση, καινούριο έλεγχο. Κυρίως πάνω στα θέματα που ακούσαμε. Όπως είπα και στην αρχή, καταλαβαίνουμε το αίτημά σας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια, θα ξεκινήσουμε αμέσως μελέτη επί των θεμάτων αυτών και όλος ιδιαίτερος θα λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που ακούστηκαν και αφορούν την Ιταλία. Ο κύριος Σλόιτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως να μην εκφράστηκα καλά, να μην υπήρξα σαφής στον πρώτο γύρο της απάντησής μου. Μακριά από μένα να διατείνομαι ότι τίποτα δεν πηγαίνει στραβά με, τους, με την κοινοτική χρηματοδότηση. Υπάρχουν ατασταλίες, Όσον αφορά την κοινωτική χρηματοδότηση και ο κύριος Φαζάκας σίγουρα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, το διαπιστώσαμε στην πρόσφατη έκθεση ε, του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας και δίνει συνέχεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναστέλουμε τις πληρωμές, άμα το επιστώνουμε αυτό, εφαρμόζουμε οικονομικές διορθώσεις και παρακολουθούμε όλες τις υποθέσεις που μας κοινοποιούνται ή κοινοποιούνται στην Όλαφ. Και βλέπουμε και τα πορίσματα της Όλαφ όταν διενεργεί έρευνε. Όταν συμπεραίνουμε τελικά ότι δεν δαπανήθηκαν σωστά τα χρήματα, ανακτώνται από εμά ή μπλοκάρονται. Έχουμε μηχανισμούς να δώσουμε συνέχεια. Όταν διαπιστώνεται παρατυπία όσον αφορά τα κοινοτικά χρήματα. Και σίγουρα θα μας ενδιέφερε να έχουμε τα σαφή ακριβή στοιχεία για ενδεχόμενες απάτες η άλλη κατάχρηση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Ιταλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να παρακολουθήσουμε και αυτά τα θέματα. Και αν έχουν διαπραχθεί απάτες πρέπει να κοινοποιηθούν στην Όλαφ. Δεν διατηνόμεθα ότι δεν πηγαίνει τίποτα στραβά, πηγαίνουν στραβά κάποια πράγματα και τα παρακολουθούμε. Αυτά και ευχαριστώ. Χαίρομαι που τελικά αισθάνεται ότι έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τη συνθήκη. Κύριε Μπαγκολή, θέλετε να συνοψίσετε, κύριε Μπεργολίτση. Ναι, γρήγορα, όπως έλεγα και πριν, είναι πολύ σημαντικός ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις νομαρχίες και με τις δικαστικές αρχές στην ε, Ιταλία, ώστε να αντισταθούμε στην, στο φαινόμενο αυτό της κακής χρήσεως των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τον οργανωμένο έγκλημα. Και θα πρέπει να αντιταχθούμε και ε, πολύ συχνά στην πλαστοπροσωπία. Πολύ συχνά οι δικαιούχες εταιρείε που παίρνουν τα χρήματα ε, είναι κάποιοι άγνωστοι, κάποιοι άνεργοι. Θα πρέπει να σταυρώνουμε τα στοιχεία και να εντοπίζουμε πραγματικά αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση. Από αυτή την πλευρά για τέτοιες επιχειρήσεις είναι σημαντικό να υπάρχει πιστοποίηση που δεν εμπλέκεται η μαφία. Θα πρέπει να αντιταχθούμε στη μεγάλη δυναμικότητα που δείχνουν οι μπρόκερ που μέσω δικτύου σχέσεων προβάλλουν, αγοράζουν ένα σχέδιο και το ξαναπολούν. Θα πρέπει να το αποθαρρύνουμε αυτό και θα πρέπει να ανοιχνεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πού πηγαίνουν τα χρήματα, την πορεία των χρημάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσω ένα παράδειγμα στην Ιταλία. Για, λόγω ενός νόμου για την ιδιωτική ζωή, αυτού που χειρίζεται την ενέργεια δεν μπορεί να κοινοποιεί τα ονόματα εκείνων που ε, ε ωφελούνται από τη χρηματοδότηση. Παίρνουν τα πράσινα ε, πιστοποιητικά. Δηλαδή προστατεύεται η ιδιωτική ζωή έτσι, αλλά είναι κάτι αντιπαραγωγικό όσον αφορά τον εντοπισμό των φορέων που θα έπρεπε να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανομαλίες. Αλλά χρειάζεται ανείχνευση των χρηματικών ροών και να πιστοποιείτε ότι ακολουθείτε η σωστή κανονική ροή. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τελειώσαμε τη συζήτηση. Όσον αφορά το σημείο αυτό τη ημερήσιας διάταξη, σίγουρα θα τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το θέμα, διότι αυτά που ακούσαμε μας δείχνουν ότι έχουμε πολλά να κάνουμε στον τομέα. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα ήθελα να πάμε στο επόμενο σημείο που είχαμε συμπεριλάβει χθε στην ημερήσια διάταξη και αφορά την απαλλαγή του Συμβουλίου. Θα ε, Μόλις μου είπαν πως ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου θα ήθελε να συμμετέχει στην ε, συζήτηση για την απαλλαγή του Συμβουλίου επίσης. Ε, θα φτάσει σε κάποια λεπτά. Α, συγγνώμη, το κατάλαβα λάθος. Θα είναι εδώ στις 11.30. 11 και 35. Θα είναι εδώ, οπότε θα διακόψουμε για να οργανώσουμε τους ομιλητές τη αποσία του κυρίου που Ladies Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε και το θέμα της συζήτηση είναι η κατάσταση πρόοδου όσον αφορά την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Στην τελευταία συνεδρίαση αρνηθήκαμε την απαλλαγή, ζητήσαμε από κάποιον να είναι εδώ από ό,τι μου είπαν απέρριψαν την πρόσκλησή μας οπότε δυστυχώς δεν είναι εδώ ο εισηγητής Είτε ο κύριος Ριβελίνη είναι στο δρόμο, έρχεται, δεν ξέρω που είναι ο κύριος Άντεργκαρντ όμως που ήταν ο προηγούμενος ε, εισηγητής μηπως μπορεί να μας πει που βρίσκεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή αν ε, μπορείτε έχετε το λόγο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς είναι μια τελείως απρόσμενη κατάσταση. Το Συμβούλιο απέριψε την πρότασή μας, την πρόσκλησή μας. Είναι μια κατάσταση βέβαια που έχει επαναληφθεί και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε παρόλα αυτά μια λύση. Η θέση μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν σαφής. Εάν δώσουμε την απαλλαγή στο Συμβούλιο, έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε ερωτήματα για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στον Ευρωπαίο φορολογούμενο δίνοντας την απαλλαγή στο Συμβούλιο χωρίς να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τους λογαριασμούς του ίδιου του Συμβουλίου. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων που θέλουμε να θέσουμε για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου. Διάφορα μυστήρια αδιαφανή και που μπορεί να εξηγούνται και που πιθανότατα δεν θα είναι προβληματικές υποθέσεις. Δεν έχουν παρά να απαντήσουν στην ερώτηση. Το πρόβλημα είναι πως δεν θέλουν να μας απαντήσουν. Και γι' αυτό το λόγο είναι ένα είδος ε, συνεννόησης με το Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει εμείς να φερθούμε. Τα δύο τελευταία χρόνια για το χρήση του 2007 και του 2008 τον, για τους λογαριασμού του Συμβουλίου υπήρχε μια, υπήρξε μια μικρή πρόοδο στην θέση του Συμβουλίου, το οποίο δέχτηκε τελικά να μας συναντήσει. Είπανε ναι, αποφάσισαν για μια άτυπη συνεδρίαση, ακόμα και αν υπήρχαν μεταφραστές διερμηνείς, αλλά έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι άτυπο, άτυπη συνάντηση. Και το Συμβούλιο απάντησε. Δεν απάντησε άμεσα, αλλά έστειλε τις απαντήσεις στην Κορεπέρ. Και η Κορεπέρ απάντησε στις ερωτήσεις μας. Και αυτές οι ερωτήσεις στη συνέχεια στάλθηκαν στο Κοινοβούλιο. Υπήρξε λοιπόν μια κάποια πρόοδος. Μα τώρα φαίνεται ότι το Συμβούλιο κάνει όπισθεν γιατί όσα είχαμε πετύχει στο παρελθόν, ακόμα και αυτές οι έμεσες απαντήσεις με εξαφανίστησαν. Αυτή τη φορά δεν λάβαμε απολύτως τίποτα και το Συμβούλιο έχει αναπτύξει νέα επιχειρηματολογία που ξεκινά από την αρχή ότι δώσαμε την απαλλαγή στην Κομισιόν και άρα αυτόματα δίνουμε και την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Δηλαδή η απαλλαγή προς την Κομισιόν καλύπτει την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να θέσουμε λέει ερωτήσεις. Και γι' αυτό και συμβουλεύθηκαν το το... συμβουλευθήκαμε τον νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Μας είπαν δεν στέκει αυτή η θέση. Δεν σημαίνει ότι επειδή δώσαμε την απαλλαγή στο Κομισιόν δίνουμε αυτόματα την απαλλαγή και στο Συμβούλιο. Είναι δύο διαφορετικά Τώρα ποια είναι τα επόμενα στάδια. Η Κομισιόν πρέπει τώρα να, ε, πάρει, να εκφράσει τη γνώμη της για την κατάσταση. Γιατί είχαν πει ότι ε, στο σημείο εκκίνησης αν ο, ή ο όρος για να δοθεί απαλλαγή προς το Συμβούλιο, αντιστοιχούσε στην απαλλαγή και στο Συμβούλιο. Αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να συμμετέχει το Συμβούλιο στην απαλλαγή του Κομισιόν. Και άρα θα πρέπει να θέσουμε τις ερωτήσεις μας στην Κομισιόν. Αλλά αυτό δεν ισχύει από ό,τι είπε η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Να μας πει και η Κομισιόν τι πιστεύει. Πιστεύει ότι το ότι δίνουμε απαλλαγή στην Κομισιόν σημαίνει και ότι δίνουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε νέες διαπραγματεύσεις για την απαλλαγή. Τέλος. Να πούμε ότι είναι αξιοθρύνητη η κατάσταση. Είναι, είναι πραγματικά λυπηρό που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή μας στο Συμβούλιο. Θα πρέπει αυτό να το παρουσιάσουμε στο σύνολο του Κοινοβουλίου, να ζητήσουμε μία, δι θέση από την Κομισιόν και να τους πούμε ότι δεν θα δώσουμε απαλλαγή παρά μόνο αν θα έχουμε ξεκάθαρη στάση και από το Συμβούλιο και από το Κομισιόν και μετά θα δούμε από τη στιγμή δηλαδή που θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ σαφή εισαγωγή. Νομίζω ότι δεν έχω τίποτα να προσθέσω διότι ε, συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι επίσης ένα θεσμικό όργανο. Πάντοτε δώσαμε απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου το Κοινοβούλιο βρίσκεται ε, ε, πλήρως νομιμοποιημένος να θεωρήσει την ε, θετική ή αρνητική άποψη του Συμβουλίου και να θα ακούσω τις απόψεις των Ευρωβουλευτών. Η κυρία Γκρέσλε. Ποτέ δεν έχω ακούσει τέτοια ανοησία σαν αυτή τη δήλωση του Συμβουλίου ότι το Συμβούλιο είναι μέρος της Επιτροπής. Δηλαδή ε, αυτό κατακριμνίζει και τη θέση του Συμβουλίου. Εάν ε, όντως το ε, αναφέρει σοβαρά αυτό το Συμβούλιο πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή και ε, να την ερωτήσουμε αν αυτή η, η συζήτηση η δήλωση ευσταθή. Αλλά τότε δημιουργείται μία κλιμάκωση του θέματος και γι' αυτό θα ήθελα το Συμβούλιο να ξανασκεφτεί την θέση του ο κύριος Κάιγερ. Στην προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει επί του θέματος είχα πει ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για ε, το θεσμικό αυτό οργανό να ακολουθήσουμε την οδό η οποία διαγράφεται διότι η συνθήκη ρυθμίζει το θέμα της απαλλαγής δεν ρυθμίζει ρητός το θέμα της απαλλαγής άλλων θεσμικών οργάνων εμείς αναλαμβάνουμε το δικαίωμα της απαλλαγής των θεσμικών οργάνων από την γενική ε, ρύθμιση Τη της απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διευκρινίζοντας και εμβαθύνοντας τις ρυθμίσεις που ήδη υπάρχουν. Πρέπει να συζητήσουμε το Συμβούλιο όπως τουλάχιστον για τα χρήματα τα οποία παίρνει από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό και ε, πρόκειται για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου αλλά καταλήγω και εγώ στη θέση την οποία και εσύ ανέφερες λέγει στην κυρία Γκλέρς λέει ο κύριος Γκάιε ε, πρέπει να ξεκινήσουμε ε, και να τους πούμε ότι είστε υπόλεγοι προς εμάς σαν εκπροσώπους των πολιτών πως εσείς εκπεραιώνετε τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές υποθέσεις. Και γι' αυτό ο, συμβουλεύω να σταθούμε ένα λεπτό και να ξανασκεφτούμε διότι η συνθήκη είναι αυτή που είναι και τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Ε, θα πρέπει όμως τότε το Συμβούλιο να μας ενάγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει ε, μία νομική γνωμοδότηση η οποία το προτείνει στο Συμβούλιο ή το υπονοεί ε, ή το συμβουλεύει και τότε μπορούν να συμβούν δύο πράγματα είτε μπορεί ε, να κερδίσουμε οπότε θα πληρώσω τη σαμπάνια ή μπορεί ε, να βασιστεί ε, το δικαστήριο εις την ισχύουσα συνθήκη και να πει ότι δεν είναι υποχρεωτικό να απαλλάξουμε το Συμβούλιο και ε, στην περίπτωση αυτή θα ε, είναι μειονεκτική απόφαση για μας αλλά ε, θα πρόκειται απλώς για μια δυσάρεστη απόφαση και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη συνθήκη μετά. Λοιπόν, εφόσον ε, ε, το θέμα είναι αν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή την ακραία κατάσταση. Διότι εγώ όσον αφορά τη δημόσια γνώμη πάντοτε μπορώ να παρουσιάσω την ε, θέση μου και να εξηγήσω ότι σαν εκπρόσωποι των πολιτών ζητώ από το Συμβούλιο να είναι υπόλογο. Και έτσι εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα εις ε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αυτό, αλλά δεδομένη της καταστάσεως αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει μέχρι την απόφαση της Ολομελίας στο τέλος του μηνός για να υπάρχει μια επικοδομητική ε, πορεία αυτού του θέματος διότι ε, ε, πιστεύω ότι δεν μας διευκολύνει το Συμβούλιο αλλά μας έχει κάνει μία προσφορά διαπραγματευτική και ο εκπρόσωπος της Ουγγαρίας είχε πει ότι ε, δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρξει ε, αλλαγή της θέσεως του Συμβουλίου αν δεν καταρτιστεί μία διαπραγματευτική επιτροπή. Δεν ξέρω ε, τι θα γίνει από αυτού, διότι έχουμε συγγράψει μία επιτολή, η οποία συζητήθηκε στους συντονιστές και όπου ρωτούμε τι θα είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και δεν ξέρω αν εσύ έχεις λάβει κάποια απάντηση αλλά το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το διαθεσμικό οικοδόμικα γιατί ε, δεν ξέρω θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις τι μέλη γενέστε. Ευχαριστώ. Εν μεταξύ ο εισηγητής έφτασε ο κύριος Ριβελίνη. Μήπως θέλετε κάτι να σχολιάσετε επί του θέματος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι έπρεπε να διανύσουμε ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο και ότι αντιμετωπίσαμε ένα δύσκολο στοιχείο. Το σύνολο της Κομισιόν και οι συντονιστές αυτούς τους μήνες, γιατί μιλάμε πια για μήνες, βρήκαν σωστό να προχωρήσουμε σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Και η θέση μας σε αυτό το διάστημα ήταν παρότι δεχόμαστε συζητήσεις από πλευράς του Συμβουλίου μάλλον εμείς μάλλον προτείναμε να γίνει συζήτηση με το Συμβούλιο, εμείς βρήκαμε μπροστά μας ένα Συμβούλιο το οποίο αγνοεί τις προσκλήσεις του Κοινοβουλίου. Όλοι γνωρίζαμε ποια ήταν τα επόμενα στοιχεία που θα μπορούσαν να... οι καταστάσεις μάλλον που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Γνωρίζαμε ποια ήταν η θέση του Συμβουλίου και των Προεδριών, Πολωνία και Ουγγαρία. Γνωρίζαμε λοιπόν ποια ήταν η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τι έπρεπε να κάνουμε. Το νέο τώρα, που δεν είναι και τόσο νέο, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου που απειλεί να προσφύγει σε άλλα θεσμικά όργανα, εύκολα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Και άρα αναλύθηκε και από πλευρά μα αυτή η περίπτωση. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλο οδός για την τιμή του Κοινοβουλίου και της ε, Επιτροπής παρά να συνεχίσουμε όπως κάνουμε εδώ και μήνες να δείξουμε δηλαδή διαθεσιμότητα για συζήτηση, γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε εμείς να συζητήσουμε. Δεν νομίζω λοιπόν πως υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, γιατί ενδεχόμενη υποχώρηση σε αυτή τη φάση θα είναι σοβαρή. Και θα είναι σοβαρή για το κύρος του Κοινοβουλίου μας. Φυσικά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους μας να φτάσουμε σε ικανοποιητική λύση. Και εγώ σήμερα το πρωί θα ήθελα στους συναδέλφους της Επιτροπής να προτείνω μια ιδέα που βεβαίω είναι προ συζήτηση θα τη θέσω. Δηλαδή να στείλουμε μια επιστολή στην ε, Κομισιόν ρωτώντας αν όντω είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη, την πολιτική και την λογιστική για τις δαπάνες που, στις οποίες προβαίνουν άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και αν είναι σε θέση να τη αρνηθούμε το δικαίωμα της απαλλαγής για ισολογισμούς που δεν έχει εκτελέσει η ίδια και οι γενικές διευθύνσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τρόπο για να ξαναπροκαλέσουμε μια συζήτηση και για να καταλάβουμε αν από την άλλη πλευρά υπάρχει βούληση αναγνώρισης των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Γιατί διαφορετικά, εγώ πραγματικά βλέπω να είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και να μην μπορούμε να κάνουμε κανένα βήμα πίσω. Μάλιστα. Η κυρία Γκρέσλε. Ε, θέλω να πω στον συνάδελφο Γκάιερ ότι μία σύμβαση μπορεί να ε, ρυθμίσει ό,τι χρειαζόμαστε καθημερινά διότι έχουμε συμφωνήσει τόσους ε, οδηγίες σε συναλλαγή με το Συμβούλιο έχουμε τα, τους διάφορους οργανισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο οπότε πιστεύω ότι μέχρι στιγμής ε, το Κοινοβούλιο είχε ένα διαμφισβήτητο δικαίωμα ελέγχου του προϋπολογισμού. Οπότε εάν το Συμβούλιο ε, ε, καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακόμη και αν κερδίσει η κατάσταση αυτή θα γίνει πολύ κρίσιμη για το Συμβούλιο Κοινοβούλιο διότι δημοσιονομική αρχή είναι το Κοινοβούλιο και αυτό προϋποθέτει ότι καταρχάς θα έχει κερδίσει και την ε, προσφυγή στο δικαστήριο. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι είναι ε, σωστό, σωστή αξιολόγησή μου ότι θέλουμε να προχωρήσουμε όπως και στο παρελθόν και να δώσουμε απαλλαγή σε κάθε θεσμικό όργανο χωριστά και αν αυτό δεν είναι δυνατόν και η συνθήκη μας, αφαιρέσει, μας αφαιρεί κάποιο δικαίωμα που είχαμε δεν ε, θα, δεν θα αποφασίσουμε αν δεν προχωρήσουμε εις ε, την ε, συνθήκη ή στην ψηφοφορία ή στην Ολομέλεια τέλος Οκτωβρίου θα δούμε τι, εάν εκεί θα ψηφιστεί η απαλλαγή του Συμβουλίου. Αν όχι θα παραπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε μετά το τέλος Οκτωβρίου τι μέλη γενέστε. Εν τω μεταξύ θα θα στείλουμε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τους ρωτήσουμε ποια είναι η θέση του. Αυτή είναι η, ε, ε, αυτό είναι το σωστό συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Συμπεραίνω λοιπόν ότι δέχεστε τα σχόλιά μου και θέλω να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου ε, στην Επιτροπή αυτή. Εδώ είναι, έχουμε τον Γενικό μας Γραμματέα, ο οποίος δεν αρνήθηκε να έρθει και θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα παράδειγμα ε, για το Συμβούλιο διότι ίσως και ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου θα ήθελε να σχολιάσει τη θέση του Συμβουλίου αλλά πρώτα θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή αν θέλει κάτι να πει και μετά θα δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα που ήρθατε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τη συνέχεια της έκθεση ε, για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου. Εγώ θα προβώ γρήγορα στα σχόλιά μου γιατί έχουμε μόνο μία ώρα στη διαθεσή μας και φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι ερωτήσει. Καταρχήν η ασφάλεια ήταν ένα μεγάλο ζήτημα ε, για αυτήν εδώ την έκθεση μετά από τα διάφορα που έγιναν εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά επίσης τα όσα συνέβησαν στις 19 Σεπτεμβρίου το blackout, τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τη γενική διακοπή δηλαδή, όπου χρειάστηκε να διακόψουμε τις συνεδριάσεις μας και να κυρώσουμε μισή μέρα δουλειάς και όπου τα πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας ε, διαφωτίσετε όσον αφορά την ασφάλεια. Επίσης, ομάδες επισκεφτών, οι οποίες ε, δημιουργούν κάποιες δυσκολίες για την διεξαγωγή των κανονικών των, των Ευρωβουλευτών. Δεν έχουμε λάβει απαντήσει εδώ. Θα μπορούσατε επίσης να μας ενημερώσετε για το πού βρίσκονται τα πράγματα και έχουμε και το λεπτό ζήτημα της πρόσβασης των Ευρωβουλευτών στο ελεγκτικές εκθέσεις ελέγχου στο ίντερνετ. Είναι δυνατόν να διατίθεται οι εκθέσεις στα μέλη, φυσικά υπό συγκεκριμένου όρου. Και αυτό θα θέλαμε να μας το απαντήσετε και έπειτα εφαρμογή του νέου καταστατικού, του νέου καθεστώτος του Ευρωβουλευτή. Επίσης ζητήθηκε αναδίπλωση επιπλέον προσωπικού καθώς και ένα πρόγραμμα δράσης και εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων. Εξεκολουθούμε να έχουμε και το θέμα των τιμών συγγνώμη, τα διάφορα βραβεία, με συγχωρείτε, ε, δεν καταλάβαμε ακριβώς, α πούμε, αυτό το τελευταίο βραβείο δημοσιογραφίας. Δεν έχουμε καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Να θίξω και ένα ακόμα θέμα. Μιλάτε για μαθήματα κατάρτιση για του ευρωβουλευτέ. Από ό,τι είχα καταλάβει, είχαμε ένα πρόβλημα. Πρόκειται για ε, κατάρτιση εβδομαδιαία που διαρκεί δύο-τρεις εβδομάδες το μήνα, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε εβδομάδα, γιατί οι δάσκαλοι δεν μπορούν να το κάνουν κάθε εβδομάδα. Είναι καλό και για τους δάσκαλους και για τους ευρωβουλευτές. Δεν ξέρω τι είδους κανόνες είναι αυτοί για τους οποίους δεν μπορούν να διδάσκουν κάθε εβδομάδα. Still, ευχαριστώ. Εδώ αυτές οι απαντήσεις είναι οι ερωτήσει, μάλλον είναι αυτές επί των οποίων θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν αρχίσουμε τη γενική ζήτηση δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. ευχαριστώ. Αυτή η άσκηση γίνεται για πρώτη φορά, διότι συνήθως ο Γενικός Γραμματέας ερχόταν μία φορά το χρόνο τον Ιανουάριο, ενώ τώρα έχουμε δύο φορές το χρόνο για να έχουμε μία γρήγορη ενημέρωση σχετικά με, τα, ε, με το ψήφισμα της απαλλαγής η οποία ψηφίστηκε το Μάιο. Σε ορισμένα λοιπόν θέμα μπορώ να αναφερθώ στην εφαρμογή, ενώ σε άλλα σημεία, εάν έχουμε έχουμε επαρκή χρόνο θα, επανέρθω, θα ε, ε, αναφερθώ σε αυτά διαφορετικά τον Ιανουάριο. Ε, θέλω να παρουσιάσω λοιπόν διάφορα από τα θέματα στα οποία πιστεύω ότι όντως έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το ψήφισμα και καταρχήν πρόκειται για τις κρίσιμες δράσεις που ενδιέφεραν ιδιαίτερο στην Επιτροπή σας οι οποίες από 88 μειώθηκαν σε 68 και δεν υπάρχει καμία μη κρίσιμη δραστηριότητα ενώ στο παρελθόν υπήρχαν τέσσερις τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δεν είχαν εφαρμοστεί ενώ εχθές μου ελέγχθη ότι τώρα δεν εκρεμεί καμία κρίσιμη ε, δραστηριότητα ε, πλέον και όσον αφορά την ασφάλεια γενικότερα. Ε, γνωρίζετε ιδίω ότι εφέτος ε, η διαπίστευση γίνεται εσωτερικά διότι χρειαζόμαστε ε, άτομα τα οποία να είναι πιστά στην οργάνωση και γνωρίζουν τους ευρωβουλευτές και έχει αλλάξει και η δημοσιονομική ε, ε, πολιτική για το 2012 και θα έχουμε εσωτερική ανάληψη ορισμένων έργων τα οποία αναθέταμε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Θέλουμε λοιπόν να ελέγχουμε όλες τις εποπτείες με το εσωτερικό μας προσωπικό. Επίσης κάναμε ε, μία αναθεώρηση όλων ε, των μηχανημάτων κάμερες δηλαδή που έχουμε για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Αποφασίσαμε να υπάρξει μία ε, νέα ε, αρχή της ε, ασφαλείας τον Ιούλιο και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πέντε διαρθρωτικές διαφορές για τον τρόπο τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε και αυτόν τον οποίο χρησιμοποιούν άλλα θεσμικά θεσμικά όργανα το ένα είναι να χρησιμοποιούμε εσωτερικό δυναμικό αντί υπεργολαβία. Επίσης ότι δεν έχουμε διάφορες ζώνες ασφαλείας. Τρίτον υπάρχει στενή συνεργασία με την τοπική αστυνομία και είναι ίσως ο πιο εμφανές σε εθνικούς οργανισμούς και δεν υπήρχε εδώ και ε, δεν έχουν καταστήματα μέσα στο κοινοβούλιο τα οποία εμείς έχουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε. Αλλά ε, όσον αφορά τις ζώνες ασφαλείας θέλουμε ε, να καταρτήσουμε σε ορισμένες περιοχές ε, ειδικέ ζώνες ασφαλείας σε συνεργασία με την Βελγική αστυνομία. Επίσης ε, υπάρχουν όλοι ε, οι υπάροχοι πληροφοριών οι οποίοι ε, είναι εντός του Κοινοβουλίου να τύχουν νέας αξιολογήσεως για να μπορέσουμε να έχουμε τα συμπεράσματα πριν από το τέλος του χρόνου με στόχο ότι ορισμένοι ε, από αυτούς τους παρόχους θα χρειαστεί πλέον να λειτουργούν εκτός της οργανώσεώς μας. Επιπλέον ε, ε, έχουμε οργανώσει τέσσερις γενικές διευθύνσεις στην αρχή τώρα έχουμε επεκταθεί σε νέα. Και έχουμε σε κάθε γενική διεύθυνση κάποια κέντρα αρμοδιότητων για θέματα προσωπικού, οικονομικά, πληροφορική κλπ και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πιο επαγγελματική αντιμετώπιση και ε, από ό,τι στο παρελθόν. Και τέλος ε, ένα μήνυμα που ίσως ενδιαφέρει το, το κέντρο επισκεπτών, το Παρλαμεντάριο και ε, ξεκινά σήμερα, ανοίγει σήμερα διότι ε, είχα σαν γενικός γραμματέας να απαντώ στο ερώτημα του πότε πρόκειται να ανοίξει το κέντρο αυτό. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σήμερα άνοιξε για το κοινό θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου και όσον αφορά τη δικιά σας άποψη για την χρησιμότητα αυτού του κέντρου ε, εγώ το επισκέφτηκα πριν 10 μέρες και πιστεύω ότι από τον 19ο το αιώνα θα προχωρήσουμε στον 21ο. Θα θέλω όμως να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη. Πιστεύω ότι είναι μια καλή επένδυση που ξεπέρασε λίγο στον προϋπολογισμό ε, και στις εκθέσεις σας ε, ζητάτε να αξιολογήσετε το διορθωτικό προϋπολογισμό και τις γλώσσες και πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού ε, έχει δεχθεί κατόπιν προτάσεώς μου ε, σε μείωση του προϋπολογισμού διερμηνίας σε 10, 10 εκατομμυρίων για το επόμενο έτος και 11 εκατομμυρίων για τη μετάφραση και με το να τελειώνουν οι συνεδριάσεις τους πιο νωρίς θα έχουμε σημαντική οικονομία και αν ε, ε, ε, έχουμε από τρίτη έως πέμπτη και όχι μόνο το τετάρτη και πέμπτη συζητήσεις θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες οικονομίες και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα απτό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποφασίσαμε με την Επιτροπή Επιτροπή Προπολογισμού ότι ε, δεν ε, θα υπάρχει μετάφραση γραπτή σε όλες τις γλώσσες, ε, θα υπάρχει μία γλώσσα και όποιος θέλει στη γλώσσα του και το ζητά θα μπορεί να του παράσχεται και η εξοικονόμηση θα είναι 8,6 εκατομμύρια. Βεβαίως επιπλέον θα μπορέσουμε με τις διάφορες διάφορες ε, άλλες ρυθμίσεις μεταφράσεως να φτάσουμε στα 11 εκατομμύρια εξοικονόμησης με τα 10 της διερμηνίας έχουμε 21 ε, και ε, με τις επιπλέον ρυθμίσεις 25,1 εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση. Ζήτατε λοιπόν καλύτερα οργάνωση. Δεν παρουσιάσαμε ένα σφαιρικό πρόγραμμα αλλά συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ήδη από το 2012. Αποφασίσαμε λοιπόν να υπάρξει και ένα πρόγραμμα για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Έχουμε περισσότερα τώρα ποδήλατα στο Στρασβούργο κατόπιν της προτάσεως που μου είχε γίνει την προηγούμενη φορά και έχουμε ρυθμίσεις με μαζικής μεταφοράς ιδίω το τρένο στο Βέλγιο για να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές διοξιδίου. Όσον αφορά τα θέματα που είχε θέσει ο εισηγητής για την ασφάλεια, νομίζω ότι έχω γενικώ απαντήσει, διότι το τελευταίο περιστατικό δεν ήταν περιστατικό ασφαλείας, ήταν ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν μπορούμε να λειτουργήσουμε όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα αλλά δεν υπήρχε κανένα κίνδυνος για κανέναν. Ε, υπάρχει όμως πρόβλημα με την επικοινωνία όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό, γιατί αν δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα ε, δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσετε και το, ε, το Προεδρείο θα το συζητήσει την Πέμπτη και επίσης υπάρχει η έκκληση να μειώσουμε τον αριθμό των επισκεφτών αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι έχοντας τώρα το πρόγραμμα το κτίριο των επισκεπτών και το 2014 με μια νέα ρύθμιση ε, θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μαζί με άλλες προβλέψεις ε, τις δυνατότητες οι ομάδες επισκεπτών να μην εισέρχονται σαν ομάδες επισκεπτών ή στο κεντρικό κτίριο θα επισκέπτονται το κτίριο των επισκεπτών το Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας και θα πρέπει να προβλέψουμε να υπάρχουν και καφετέριες, εστιατόρια αλλά με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική μπορούμε να οργανώσουμε το κέντρο κέντρο επισκεπτών μας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην κατακλείζουν οι επισκέπτες αυτές τους διαδρόμους, τα σανσέρ και να μας δυσχεραίνουν τη ζωή. Ε, επίσης ε, μας είπατε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού ε, θα συζητούσε ορισμένα θέματα μαζί μας. Μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει. Ίσως αυτό οφείλει στο ότι αλλάξατε πρόεδρο και είμαι βέβαιος ότι ο νέος πρόεδρος θα με προσεγγίσει επί του θέματος και θα το συζητήσουμε. Θα υπάρξει και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού η οποία είναι εν εξελίξη και είμαι στη διάθεση ε, του Προέδρου να το συζητήσουμε όποτε επιθυμεί. Για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού ε, έχουμε δύο θετικές αξιολογήσεις στις γενικές Γενικής Διεύθυνσης ε, Οικονομικών αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε τις αντιδράσεις των υπευθύνων ε, οργανισμών και πρώτα απ' όλα του Προεδρείου το οποίο ε, θα πρέπει να μας δώσει την άποψή του και όταν το Προεδρείο έχει ολοκληρώσει την εξέταση και τη συζήτηση θα έχουμε τα συμπεράσματα αλλά δεν μπορούμε χωρίς αυτές τις εκθέσεις να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συστάσεις. Ε, όσον αφορά τις τιμές, μέχρι στιγμής το Προεδρείο δεν έχει αναθεωρήσει την άποψή του για τις τιμές σχετικά με τα ε, ε, εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει να δούμε αν οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι έχουν διαφορετικές ανάγκες και να προσαρμοστούμε, αλλά έχω κάνει μία πρώτη εισαγωγή και μία μία πρώτη παρουσίαση και είμαι στη διάθεσή σας για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. κύριο Σίταλα θέλει να πει κάτι. Δεν αναφέρθηκα στην ε, πολιτική των κτηρίων γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω αργότερα να επανέλθω λοιπόν στο θέμα των κτηρίων, της πολιτικής των κτηρίων. Καλώς. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Και ο Σχερ Μπράντι είναι ο πρώτος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χθες το πρωί έφτιαξα καφεδάκι. Και αποφάσισα να διαβάσω το έγγραφο πίνοντας τον καφέ. Που λάβαμε τον κύριο Βέλε. Γιατί το λέω αυτό. Ήρθα να περιγράψω ότι ήταν καλή η διάθεσή μου. Έξω έβρεχε. Άρα δεν είχα αντιπερισπασμό και μπορούσα να συγκεντρωθώ στο έγγραφο. Άλλαξε όμως τη διάθεσή μου διαβάζοντας το έγγραφο. Να προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί. Εξεπλάγει από τον τόνο του εγγράφου πολύ. Στα μισά δεν ήμουν σίγουρα στη διάβαζα διάβαζα νέο σενάριο σειρά του BBC, το νέο μάλιστα κύριε Υπουργέ, ή σοβαρή απάντηση στην επιστολή, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Με εξέπληξε ο τόνος του κειμένου. Να δώσω κάποια παραδείγματα στον αφορά το ύφος του κειμένου. Ζητήσαμε κάτι να γίνει όσον αφορά το βραβείο δημοσιογραφίας και ότι διαδικασία για το βραβείο για δημοσιογραφία του 2011 ξεκίνησε πριν από την αθέτηση του εν λόγω ψηφίσματος. Γιατί είμαστε πιο δραστήριοι, να πούμε ότι ετοιμάζουμε ένα έγγραφο συζήτηση για το Προεδρείο, να συζητηθεί το μέλλον του ε, βραβείου για τη δημοσιογραφία. Βάζουμε τα υπέρ και τα κατά για να συνεχιστεί η συζήτηση από αυτού και άλλων συναφών θεμάτων για το τι γίνεται με τα αμοιβή των ε, ντόπιων βοηθών και τα τιμολόγια. Είπατε ότι μπορούν να πληρωθούν τιμολόγια εντό τριών εβδομάδων αν συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο και ε, προ, ε, καταβληθούν εντός των προθεσμιών. Ε, όμως εξακολουθούν να καταβάλουν τιμολόγια τώρα χωρίς να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Και γι' αυτό τελικά γίνονται, υπάρχουν καθυστερήσεις σε αυτή την πληρωμή. Μα εδώ είναι η καρδιά του προβλήματος. Ίσως δεν είναι το πρόβλημα που δεν ακολουθούμε τους κανόνες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να προστεύσουμε τους κανόνες. Άλλο ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Για το γραφείο ταξιδίων, για φθηνότερες πτήσεις. Λέει ότι το σύστημα κρατήσεων αμεντέους ε, δεν έχει τις φθηνότερες αεροπορικές εταιρείε. Γιατί όχι. Γιατί να μην μπούμε να βρούμε τρόπους να συμπεριλάβουμε τις φθηνές εταιρείε um, στο σύστημά μας για τα μίλια αεροπορικών ταξιδιών. Περιγράφεται το πώς δύσκολο είναι ότι δεν γνωρίζετε πόσα μίλια κάθε βουλευτής συλλέγει κλπ. Βεβαίως όχι, αυτό είναι ένα θέμα του προβλήματος. Γιατί να μην πούμε καλό, το εξετάζουμε, Ήρθαμε σε επαφή με το Δανέζικο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, διότι ήδη έχουν αυτό το σύστημα. Οι εθνικοί βουλευτές χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους μίλια για τις επόμενες πτήσεις τους. Πού υπάρχει η ενεργής, η ενεργός διάθεση για βελτίωση. και δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου. Αυτή η νοοτροπία, αυτή η στάση, πώς βλέπετε το ρόλο σας. Εξετάζοντας το ψήφισμα και προσπαθώντας να μας βοηθήσετε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αντί να το κάνετε αυτό, τι πιστεύετε, πιστεύετε κάποιες ιδέες είναι καλές ή θεωρείτε ότι ρόλο σας είναι να προσπαθείτε να ελιχθείτε μέσα από τις γραμμές του ψηφίσματος και να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς να αλλάξει κάτι. Σοβαρότατο αυτό το ερώτημα. Ποια είναι η στάση σας, ποια είναι η νοοτροπία της γραμματείας. Ποια είναι η στάση της γραμματείας έναντι του προπολογισμού του Κοινοβουλίου και έναντι του ψηφίσματος της ύψης της πολιτικής αρχής του Κοινοβουλίου, που είναι η Ολομέλεια και όχι το Προεδρείο. Κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Τα μίλια ήδη τα ανέφερα. Θέλω το σχόλιο σας. Δεν αναφέρεστε καθόλου στην παράγραφο 135. Εκεί ζητάμε πιο ενεργό τρόπο για τη μείωση της ε, χαρτούρας στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια εφαρμογή για τους υπολογιστές, για τα tablets, όπου να μπαίνει σε μια θέση να πατάς ένα κουμπί και να σου έρχονται όλα τα έγγραφα στον υπολογιστή σου, στην ηλεκτρονική σου συσκευή. Πρέπει να είναι δυνατόν όμω, σαν βουλευτή, να πει ότι δεν χρειάζεσαι χαρτί. Όταν σε έναν κατάλογο για μη συνεδρία επιτροπή να μην σου δίνουν τα έγγραφα σε χαρτί. Χρειαζόμαστε τα έγγραφα βέβαια, αλλά πολύ συχνά μπαίνω σε μια αίθουσα που υπάρχει ένα βουνό, σωρό από χαρτί. Και δεν μπορώ να πω εκ των προτέρων ότι μου χρειάζεται, μου το τυπώνω έτσι κι άλλιω. Θέλω απάντηση σε αυτό, για τα ποδήλατα. Έχουμε 10 ποδήλατα στο Στρασβούργο από το Κοινοβούλιο. Είπατε ότι θα έχουμε 100 με 150 από την πόλη του Στρασβούργου. Πρώτα απ' όλα, τώρα υπάρχουν 30 ποδήλατα. Δεν δουλεύει αποτελεσματικά το σύστημα πέραν από αυτό. Εγώ θα θέλω να εξαρτώ με λιγότερο από την πόλη του Στρασβούργου. Ίσως του χρόνου να αποφασίσει στο Στρασβούργο να απαλλαγεί τα ποδήλατα γιατί είναι πολύ ακριβά και να έχουμε μόνο 10 ποδήλατα. Εγώ τι ήθελα. Όχι μόνο αυτά τα ποδήλατα, αλλά να δείξει το Κοινοβούλιο ότι δεν σκεφτόμαστε μόνο τα μεγάλα αυτοκίνητα, αλλά σκεφτόμαστε και άλλους τρόπους μεταφοράς, κυρίως σε μια πόλη σαν το Στρασβούργο, που έχει φτιαχτεί για τα ποδήλατα. Σκεφτείτε το κι αυτό. Τέλος. Πρόεδρε. Ζητήσαμε μακροπρόθεσμη αναθεώρηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Και τι οικονομίε να κάνουμε στο μέλλον ενδεχομένω. Αναφέρατε κάποιε οικονομίε. Για να είμαι ειλικρινή, από πλευρά από το 1,7 δι ευρώ, αυτά τα λίγα εκατομμύρια που αναφέρατε δεν είναι κάτι που θα μας οδηγεί σε επικεφαλίδες στον τύπο ότι προσπαθούμε να κάνουμε οικονομίες στο Κοινοβούλιο. Στον προπολογισμό του 2012 και το σχετικό ψήφισμα που θετήσαμε τον Μάιο, ζήτησα μια επισκόπηση ενδεχομένων οικονομιών, υιοθετήθηκε από τον Λομέλια, που είναι η ψηστή πολιτική αρχή, που ζήτησε από τη Γραμματεία να δώσει μια ανάλυση ενδεχομένων δυνατών οικονομιών, δεν λάβαμε τίποτα ακόμα. Το ζήτησα αυτό πριν τη διαδικασία προπολογισμού του 2012. Χάσαμε αυτή τη διαδικασία, ίσως για του χρόνου μπορείτε να μας το διαθέσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά εισαγωγικά ερωτήματα, καλό ερώτημα. Αλλά αν όλοι χρειαστούν το ίδιο χρονικό διάστημα, όλοι που έχουμε στον κατάλογο, θα τελειώσουμε περίπου στις μισή. Προτείνω λοιπόν, αν επιτρέπετε, πόσους έχω στον κατάλογο, έχω άλλους έξι ομιλητές. Προτείνω λοιπόν να περιοριστούμε στο δίλεπτο ο καθένας. Λυπούμε που δεν είχα τη δυνατότητα να το πω για τον πρώτο μιλητή, το λέω τώρα και μετά ο Γενικός Γραμματέας θα απαντήσει στι ερωτήσει. Άλλο θέλει να μιλήσει στον κατάλογο εσεί. Κάποιος που δεν σήκωσε το χέρι του και θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, ορίστε. Κλείνουμε τον κατάλογο. Ο κύριος Έπινγκ λοιπόν έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, πιο σύντομος από τον συνάδελφό μου. Πρέπει να παραδεχτώ ότι πολύ συχνά δεν συμφωνώ μαζί του, σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ. Άρα μπορώ να συνεχίσω. Αύριο δημιουργείται ομάδα προβληματισμού του ECR που θα παρουσιάσει, παρουσιάσει έκθεση. Τέλος της υπερβολής και θα αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να μειώσουμε κατά 24% τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Νομίζουμε ότι είναι δυνατόν. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα μικροπράγματα, τα ψίχουλα, όπως έκανε ο ο Βέλερ, αλλά τις δομικές, τους δομικά αίτια. Ο κ. Στάς είχε κάνει σωστή ανάλυση. Δυστυχώς δεν είναι εδώ για να υποστηρίξει το σχόλιο μου αυτό. Και ποια ήταν τα συμπεράσματά του. Συμπέρασμα. Βλέποντα τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι βλέπει, τεράστια αύξηση τη γραφειοκρατία. Έχουμε ένα κύμα γραφειοκρατία στη Γερμανία. σε βέλε θα το λέγαμε. Δεν θέλω να συνδέσω αυτό με, τα, με το Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Το 2004 ο αριθμός υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκε από 4.000 σε πάνω από 6.200. 6.200 ευρώ βουλευτές αυξήθηκαν μόνο ε, κατά τέσσερις. Από πού προέρχεται όλο αυτό το πλεόνασμα. Η διαδικασία ε, οδηγείται από τη γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε διαθροτικές περικοπές. Και αύριο θα παρουσιάσουμε την έκθεση και θα στείλω και αντίγραφο στον κύριο Ζητής... Υποβάλαμε 20-30 ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο Χρειάστηκε τρίμηνο το Κοινοβούλιο να απαντήσει στις μισές. Όμως είχαμε τουλάχιστον επαρκείς πληροφορίες για να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε περικοπές στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να περικόψουμε 400 εκατομμύρια και να δείξουμε ότι όταν οι πολίτες περνάνε μια κρίση, εμείς δεν μπορούμε να τα γνώμε. Νομίζω ότι πέρασε το δίλεπτο, λέει ο Πρόεδρος, παρακαλώ ολοκληρώστε. Κύριε Έπινγκ, θα υποβάλουμε την έκθεσή μας στον κύριο Βέλε και θα τον βοηθήσουμε να σκεφτεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ε, κυρία Κρέσλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι ε, έχουν γίνει ε, πρόοδοι γιατί είμαι παλιό μέλος και ξέρω πόσο δύσκολα ήταν η κατάσταση προηγουμένως. Βλέπουμε ότι τώρα ε, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε τσακωθεί επί χρόνια με τη διαχείριση και δεν είναι η κατάσταση όπως την παρουσιάζει ο κύριος Γκέρ Μπράντι διότι ε, έχουμε μία έκθεση κατά πρωτοβουλία σχετικά με το γλωσσικό θέμα και ελπίζω ότι μπορούμε να προετοιμάσουμε την επόμενη φάση. Πού ήσασταν αγαπητοί συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια, διότι είχα ζητήσει ε, πάρα πολύ καιρό τώρα να υπάρχει ε, μία εξέταση, ένα screening του ε, προσωπικού του Κοινοβουλίου όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γι' αυτό και χαιρετίζω τις εξελίσεις που έχουν γίνει. Ε, έχω όμως δύο ερωτήσεις. Καταρχήν για το Παρλαμεντάριουμ, για το κέντρο των επισκεπτών. Ακούω πολλά ωραία πράγματα και μου λένε γιατί χρειαζόμαστε και το Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πεςτε μου λοιπόν τι πρέπει να απαντήσω. Δεύτερον, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των Ευρωβουλευτών. Ε, έχω έναν τρίτο βοηθό, χρειάζομαι και ένα τηλέφωνο για αυτόν. Δηλαδή είναι θέματα που πρέπει να συντονίζουμε και καλό θα ήταν να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Διότι ε, θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα καταρτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν το ξέρουν όμως όλοι. Έχουμε πρόσβαση στην Επιτροπή στα προγράμματα αυτά. Αν ναι, καλό θα ήταν να δημοσιοποιηθεί. Ευχαριστώ κύριε Ζόντεγκατ. Ευχαριστώ. Λόγω του χρονικού περιορισμού θα συγκεντρωθώ σε αυτή τη διακοπή του ρεύματος. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η διακοπή οφειλόταν σε πυρκαγιά εκτός πόλης. Από ό,τι θυμάμαι, έγινε κάποια συζήτηση που έλεγε ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα εφεδρικό στο Κοινοβούλιο ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα χρειαζόταν χρήματα αυτό το σύστημα και θα δημιουργόταν κάποια δομή, υποδομή. Όταν πατήθηκε λοιπόν το κουμπί του εφεδρικού συστήματος, τι συνέβη. Σπαταλήσαμε τα χρήματά μας, τα χάσαμε. Τι συνέβη τελικά με το εφεδρικό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ ο κύριος Όχι. Ο κύριο Γκάιερ έχει το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε ε, ε, καιρό να ακούσουμε τις αντιδράσεις της, ε, στα σχόλια του κυρίου Έπινγκ αλλά εδώ έρχομαι σε ένα θέμα που μου είναι προσφυλές την πολιτική των κτηρίων και σε αυτό το σημείο ε, με τους υπαλλήλους της Γενικής Διευθύνσεως σε συνεχή διένεξη για το θέμα των κτηρίων. Γι' αυτό και τώρα ζήτησα να υπάρξει μία ανάλυση η οποία θα μπορέσει να μας δείξει τις δαπάνες, την καταβολή κεφαλαίου, κόστος ανατετραγωνικών και πόσο συγκρίνεται από πλευράς τιμής ένα κτίριο στην σημερινή κατάσταση της αγοράς στις Βρυξέλλες διότι Πρέπει, πρέπει να μπορεί κανείς να κάνει μία σωστή αξιολόγηση και να δούμε αν είναι σωστή η στρατηγική του Κοινοβουλίου να αγοράζουμε αντί να νοικιάζουμε. Όταν τα, βλέπω λοιπόν όλα αυτά βλέπω ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη και ε, ίσως θα πρέπει να προσελκύσουμε διάφορους οργανισμούς πιο κοντά μας. Μπορείτε λοιπόν να δικιά σας σκοπιά παρακαλώ να μας κάνετε μία μελέτη η οποία θα μας βοηθήσει να κάνουμε τις συγκρίσεις. Ευχαριστώ ο Ανδρέας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα θέμα δεν θέσατε. Τα σανσέρ, τους ανελκυστήρες. Και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα δύο-τρεις ευρωβουλευτές ε, από, έπεσαν από τον πρώτο όροφο στο πρώτο υπόγειο. Είναι εξωφρενικό αυτό που συνέβη σε αυτό το κτίριο. Και στο Στρασβούργο πρέπει να τρέχουμε 10-15 λεπτά πριν από τις ψηφοφορίες διότι δεν έχουμε αρκετό χώρο στα σανσέρ κινούνται πολύ αργά. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Δεν άκουσα τίποτα πάνω σε αυτό. Άλλο ερώτημα. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο αυτή η μελέτη για το νέο καταστατικό των μελών. Μετά από ένα χρόνο πρέπει να έχουμε αυτή την αξιολόγηση. Ακούγονται παντού φήμες, σύμφωνα με τις οποίες το καταστατικό ε, αυτό το καινούριο γίνεται πιο ακριβό από το παλιό. Και κάθε φορά που πάω στο γραφείο πληρωμών βλέπω ότι η δίκηση έχει υπερφορτωθεί, ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τι περιμένουμε. Θα γίνει η μελέτη, θα την έχουμε στα χέρια μου το τέλος της θητείας αυτής ή περιμένουμε για την επόμενη. Τελευταίο ερώτημα της κυρίας Αντριάσον. Ε, γιατί χρειαζόμαστε κέντρο επισκεπτών γιατί χρειαζόμαστε το τον ευρωπαϊκό οίκο τη ιστορία ε, αυτή την εποχή τη κρίση. Αυτό είναι προπαγάνδα. Η καλύτερη προπαγάνδα για το Κοινοβούλιο θα ήταν να έχει κόσμο που ξέρει ότι υπάρχει κρίση, ότι σπαταλούν, ξοδεύουν λίγα χρήματα του φορολογούμενου και κάνουν καλή δουλειά. Να μην ε, υπάρχει όλη αυτή η προπαγάνδα. Ο κ. Μπαλσίτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτούς που επένεσαν το Γενικό Γραμματέα για τα βήματα που έκανε, που μας επιτρέπουν να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση χρημάτων και στα δυόμιση χρόνια που συμμετείχα στις διάφορες συνεδριάσεις πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την χρήση των χρημάτων. Έχω 15-20 ερωτήσεις που σημείωσα που θα μπορούσα να θέσω, αλλά νομίζω ότι βασικό στόχος σήμερα είναι να κάνουμε τις μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες χωρίς να μειώσουμε τις συνθήκες, ε, εργασίας, συνθήκες για τους βουλευτές. Ζούμε σε διάφορες χώρες και ερχόμαστε κάθε εβδομάδα από διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ποικίλουν οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά που κάνουμε. Ένα μεγάλο θέμα, νομίζω, είναι αυτό που ε, σχετίζεται με τις καντίνες, με τα εστιατόρια, την ποιότητα του φαγητού. Το είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι δεν μπορεί να λυθεί εύκολα το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε το πρόβλημα όμως. Από την άλλη, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι θα ήταν σόφρον να ε, έχουμε κάποιο είδους ε, συμβάσεις ε, για μισθώσεις και κάποιες συμβουλές για τις μισθώσεις. Για μας που ερχόμαστε στο Βέλγιο και δεν ξέρουμε το εθνικό δίκαιο και παραβιάζονται τα δικαιώματά μας θα πρέπει να έχουμε αυτές οι συμβάσεις να μας βοηθούν διερμηνία, μετά Είναι σωστή η πρόταση, είναι αποτελεσματική, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα. Αν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων να θα συμμετέχουμε ή όχι σε συνεδρίαση. Και συμφωνώ ότι για την απαλλαγή του 2010 ίσως να έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται στο θέμα αγοράς και ε, μισθώσεων ε, των κτηρίων. Κυρία Χώσμαερ. Καταρχήν ε, μία συγκεκριμένη ερώτηση για το γραφείο ταξιδίων. Το πρόβλημά μου δεν είναι το σύστημα Μαντέους, αλλά όπως και άλλοι συνάδελφοι πιστεύω ότι εάν θέλει κανείς ε, να κλείσει μία πτήση και ε, αν ε, κάνουμε την κράτηση μόνη μας είναι πολύ πιο ευνοϊκή η τιμή μέχρι χίλια ευρώ φτηνότερα και προσπάθησα επίσης να κλείσω ένα ξενοδοχείο μόνιμο ή μέσω του γραφείου ταξιδίων και είδα ότι η προσωπική μου τιμή μπορεί να ήταν μέχρι 100 ευρώ φτηνότερη και είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με αυτό το γραφείο ταξιδίων. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται μεγαλύτερες δαπάνες από το γραφείο ταξιδίων ασχέτως των αεροπορικών εταιριών. Επίσης το θέμα των οδηγών, διότι σε ορισμένα κράτη Υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι πιο ευνοϊκά. Ε, σκέφτομαι δηλαδή και τα έξοδα ταξί. Ε, το σύστημά μας πιστεύω δεν είναι πολύ αποτελεσματικό και θα ήθελα να ακούσω κάποια πρόταση. Ε, και όσον αφορά τον κύριο Γκάιερ έχουμε όντως προσπαθήσει να κάνουμε συγκρίσεις και θα δούμε ότι σε κάθε ερωτήριο ερωτηματολόγιο συγκρίνουμε το κόστος της ε, οικοδόμησης με το, της αγοράς με το κόστος της ενοικιάσεως. Δηλαδή ε, δεν ε, αγοράζουμε κανένα κτίριο αν θα ήταν ευνοϊκότερη ενοικίεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε διαπιστώσει σε κάθε φάση της συγκρίσεως αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείτε να επαληθεύσετε. Ε, όσον αφορά το κέντρο των επισκεφτών ε, και ε, αναρωτιέμαι αν δεν υπάρχει επικάλυψη με το Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας διότι ίσως δεν προγραμματίστηκαν και τα δύο την ίδια στιγμή και κατά την άλλη κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω τώρα καλύψει τον κατάλογο των ομιλητών και δίνω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ίσως ε, όσον αφορά τον κύριο Γκερμπράντι. Καταρχήν, Πιστεύω ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι λήψεως αποφάσεων στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή η Επιτροπή ε, ε, ε, ελέγχου του προπολογισμού αποφασίζει για την απαλλαγή αλλά η Επιτροπή Προπολογισμού αποφασίζει επί του προϋπολογισμού και ούτε η μία ούτε η άλλη δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του Προεδρείου. Υπάρχουν δηλαδή τρεις διαφορετικές διαδικασίες για τον προπολογισμό, για τον έλεγχο προϋπολογισμό και για τον Πρόεδρο εγώ είμαι υπεύθυνο για τη διαχείριση. Δεν μπορώ ούτε να αντικαταστήσω τους πολιτικούς υπευθύνου ή να προκαταλάβω τι θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε ότι η γλώσσα μου είναι προσεκτική. Χρειαζόμαστε αποφάσεις είτε της Ολομελίας είτε του Προεδρείου για θέματα ε, ίσως δεν άπτονται του ελέγχου προπολογισμού αλλά του προπολογισμού. Δηλαδή ο κάθε τομέας μπορεί να λάβει τις δικές του αποφάσεις. Ως προς τις αντικειμενικές ερωτήσεις, μάλλον επί συγκεκριμένων θεμάτων όσον αφορά τα μίλια στις αεροπορικές εταιρείες. Τις επαφές που είχαμε μέχρι τώρα με τις αεροπορικές εταιρείες μας είχαν πει ότι δεν ήταν έτοιμες οι αεροπορικές εταιρείες να πιστώσουν τα μίλια ή στη διοίκηση. Πρέπει όμως να το ξαναεπαληθεύσουμε στην τωρινή δημοσιονομική διαδικασία και φαντάζομαι ότι θα γίνει αποδεκτό από την Ολομέλεια διότι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος κατά 4,1 εκατομμύρια με τέσσερους τρόπους είτε να μειώσουμε το κόστος για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών μέχρι των ομιλίων πρέπει να το ελέγξουμε ε, θα δούμε την ε, Παρασκευή τι θα έχει γίνει επί του θέματος και επίσης θα μειωθεί το κόστος όχι μόνο ο ε, για ε, τους συνεργάτες αλλά για, για τους ευρωβουλευτές και η απόφαση θα ληφθεί μεταξύ Επιτροπής Προπολογισμού και Προεδρίου και βεβαίως το, η εξοικονόμηση των 4,1 εκατομμυρίων δεν είναι πουσιώδης. Επίσης όσον αφορά τα έγγραφα έχουμε ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει ε, στις επιτροπές όλα να γίνονται χωρίς έγγραφα και αυτό το δοκιμάζουμε σε δύο επιτροπές για να γενικευθεί το πρόγραμμα αυτό σε όλες ε, τις επιτροπές και στο τέλος ε, της ε, θητείας αυτής θα μπορέσουμε να εγκαταλείψουμε τελείως την χρήση των εγγράφων. Να υπάρχουν λάπτοπ σε όλα τα γραφεία και ο κάθε ευρωβουλευτής να έχει μία ταμπλή ταμπλέτα. Εγώ προχώρησα σε αυτήν την λύση, δεν μου χαρίστηκε ο τύπος της Ευρώπης, αλλά μπορώ να σας πω ότι έτσι εργάζομαι πολύ καλύτερα. Όσον αφορά την εξοικονόμηση και τις οικονομίες, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε το κατά 25 εκατομμύρια και πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο ποσό που πρότεινε κάποιος γενικός γραμματέας να εξοικονομήσει. Για πολλούς δεν επαρκεί αλλά δεν πρόκειται για πενταροδεκάρες είναι ένα σημαντικό ποσό και μπορώ να σας πω ότι στο παρελθόν οι γλωσσικές υπηρεσίες δεν είχαν υποστεί περικοπές και εδώ βρισκόμαστε ε, σε ένα νέο τομέα και δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι προσπάθειες. Θα έπρεπε μάλλον να αναγνωριστούν. Για τον κύριο Έπινγκ. Ε, στην αρχή ε, είχα την ε, ίδια, το ίδιο σχόλιο είσαστε μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού ξέρετε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι αρμόδια για τα θέματα της και πρέπει να σας πω ότι το 2004 εφόσον διευρυνθήκαμε κατά δέκα κράτη ε, έχουμε ένα πλήρες γλωσσικό καθεστώς. Δηλαδή ε, σε αντίθεση με το Συμβούλιο θέλουμε να έχουμε πολυγλωσία σε όλες τις γλώσσες. Για μας αυτό σημαίνει ότι μία επιπρόσθετη γλώσσα σημαίνει 50 ε, νέου μέλη στην μετάφραση, 30 επιπλέον διερμηνείς και επιπλέον επικοινωνία ε, ε, γραφεία εξωτερικά, ε, δηλαδή μεγαλύτερες δαπάνες και καλύτερος εξοπλισμός. Χρειαζόμαστε δηλαδή τουλάχιστον 30 επιπλέον συνεργάτες και ακολουθούμε την πολιτική του Κοινοβουλίου η οποία είναι να υπάρχει πλήρης πολυγλωσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν αυτό το πολλαπλασιάστε επί 10 για τις 10 νέες χώρες σημαίνει ότι έχουμε ε, ε, επί 30 συνεργάτες πολλούς περισσότερους και αυτό δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Γκρέσλε σας μίλησε για το Μουσείο Ιστορίες. Θα πρέπει όμως ε, τις επόμενες μέρες να επισκεφθούμε το κέντρο επισκεφθών για να έχετε ίδια εικόνα. Θα δείτε όμως ότι εδώ αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μία γρήγορη ιστορική αναδρομή στα βασικά οπτικά γεγονότα, προσπαθούμε όμως με ε, οπτικά μέσα και ε, πολλαπλή μέσα να ε, δείξουμε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου που είναι τελείως διαφορετικό θέμα από την ιστορία και ιδίως την ιστορία της ενώσεως της Ευρώπης. Αυτό που είναι για μένα μία πολύ καλή εξέλιξη είναι ότι μας έγραψε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διευκρινίζει Ελπίζω το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο κόστος και ελπίζω ότι ε, για το 2013 θα έχουμε μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα αυτό διότι ε, το, το Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν αναφέρεται μόνο στο Κοινοβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα μπορούν να συμμετάσχουν. Θα έρθουν και ε, σκέπτες από το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο άρα σωστό είναι αυτή, αυτά τα έξοδα να μην τα αναλάβει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το καλοκαίρι και μετά από παρέμβαση του προεδρίου έχει μειωθεί το τρέχον έχουν κόστος κατά 20 ε, εκατομμύρια και ε, πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από το Προεδρείο επί του θέματος. Ε, Όσον αφορά τις κεντρικές λειτουργίες και ενφουξιών, δεν θυμάμαι σε τι το είχα αναφέρει, αλλά ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε διμερώς. Σχετικά με την πολιτική κτηρίων, όπως είπε η κυρία Χολμάγερ, όντως συγκρίνουμε την τιμή αγοράς και νοικιάσεως, αλλά το ουσιαστικό μας πρόβλημα είναι ότι πάντοτε και θεωρώ ότι είναι σωστό και πρέπει να επιμένουμε, τα κτίρια μας δεν πρέπει να είναι διεσπαρμένα σε όλη όλη την πόλη. Εάν μοιράσουμε τα κτίρια μας σε όλη την πόλη μπορούμε να πούμε πού υπάρχει η ε, πιο ευνοϊκή τιμή ανά τετραγωνικό αλλά αυτό έχει επιπτώσεις, δεν υπάρχει καλές συγκοινωνίες, υπάρχει κόστος μεταφοράς και προβλήματα, έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε και όλα αυτά τα θέματα διότι πάντοτε η προσφορά κτηρίων είναι περιορισμένη ε, δεν είναι καλή η διαπραγματευτική μας θέση γιατί και ο πολιτής ε, ξέρει ότι το κτίριό του είναι κοντά στο κοινοβούλιο αλλά πρέπει να σας πω τώρα ότι ε, εξετάζουμε τώρα την μεσοπρόθεσμη εφαρμογή της πολιτικής κτηρίων και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας μιλήσω ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν διότι εξετάζουμε την αγορά, τα ενίκια, τις διάφορες διαδικασίες αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε και άλλες προτάσεις στο Προεδρείο για την πολιτική κτηρίων πριν τελειώσει ο χρόνος διότι καταρχήν θέλουμε να μεταφέρουμε άλλες ε, υπηρεσίες από το κτίριο Eastman, μετά το professional training, μετά το παιδικό σταθμό των υπαλλήλων και θα χρειαστούμε επιπρόσθετα κτίρια. Η κυρία Ανδρέασεν ε, μας είπε ότι δεν απάντησα για το ασανσέρ. Ε, δεν απάντησε γιατί δεν με είχε ρωτήσει κανείς, αλλά μπορώ να σχολιάσω το θέμα αυτό. Δεν έχουμε επαρκή ασανσέρ για τον αριθμό των ατόμων στα κτίρια, διότι τα κτίρια μας προβλέπονται, ε, ε, προβλεπόντουσαν για άτομα που έχουμε υπερβεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορούμε ε, λοιπόν να εργαστούμε με αυτό τα άτομα εις τα κτίρια, γι' αυτό και αναφερθήκαμε εις τους επισκέπτες επισκέπτες, εάν θα δεχόμαστε επισκέπτες στα κτίρια μας που επιβαρύνουν ε, τα σανσέρ και τους διαδρόμους. Υπάρχει υπερβολική επιβάρηση των κτιρίων μας. Έχουμε ε, ε, ανεπαρκή και υπερβολική ε, αριθμό ατόμων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά το θέμα των επισκεφτών. Γι' αυτό και ε, θα ήθελα να υπάρχει μία αντιμετώπιση των επισκεφτών μέσω του ε, ε, κέντρου επισκεπτών του Μουσείου Ευρωπαϊκής Ιστορίας και μία επίσκεψη της Ολομελίας η οποία έχει αυτή τη δυνατότητα προσθεθεί μια έξοδος. Μετά, όσον αφορά την αξιολόγηση του καταστατικού, όσαν ε, ε, υπάρχει μια επιτροπή υπό την κυρία Ροντ Μπέρεντ, η οποία συνεχώς παρακολουθεί τις αδυναμίες της εφαρμογής του καταστατικού, τόσο για τους βοηθούς όσο και για τους ε, ευρωβουλευτές. Δηλαδή, αν αν κάποιος δεν γνωρίζει όλα τα προβλήματα δεν μπορεί να συνυπολογίσει όλες τις επιπτώσεις. Προβλέπουμε λοιπόν ε, ότι θα προχωρήσει η εργασία αυτή ακόμη δύο χρόνια αλλά τώρα πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή, να γίνει μια αξιολόγηση η οποία θα υποβληθεί στην ομάδα εργασίας και στη συνέχεια ε, στο Προεδρείο και η απόφαση θα έχει ληφθεί μέχρι τέλος του έτους ε, διότι έχει ερωτήσει πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα γίνει πριν τη μέση της θητείας του Κοινοβουλίου και ε, μπορεί ο καθένας να καταλήξει σε συμπεράσματα και εμείς ε, σαν διαχείριση, ε, σαν διαχειριστικό όργανο θα έχουμε οδηγίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλτσίτης για αυτά τα οποία αξιολόγησε, δηλαδή ότι χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο χρηστά τους πόρους μας και για τις συνθήκες ε, για τους ευρωβουλευτές που μας απασχολούν όσον αφορά το εστιατόριο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε μόνο μία μεγάλη κουζίνα και από τη μία μεγάλη κουζίνα ουσιαστικά ε, τροφοδοτούνται και όλα τα εξωτερικά ε, σημεία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Δεν μπορεί την κουζίνα αυτή να τη χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε. Πρέπει αν, αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πολλές παροχές να μην έχουμε μόνο μία κουζίνα αλλά δύο ή τρεις κουζίνες από τις οποίες ε, οι διάφοροι πάροχοι μπορούν να εργάζονται και υπάρχει ανταγωνισμός. Στο τομέα του αισθητορίου της καντίνας ε, έχουμε δύο-τρεις μεγάλους παρόχους οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μας και άρα δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Για να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός χρειαζόμαστε περισσότερους ενδιαφερομένους αλλά και περισσότερες κουζίνες για να ε, δίδονται υπηρεσίες επιτόπου. Στην αρχή θα χρειαστούμε δύο και ε, τρία μεγαλύτερα εστιατόρια τα τα οποία θα μπορούν να τροφοδοτούνται χωριστά, οπότε ε, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για την ένδειξή σας για τις γλωσσικές υπηρεσίες on demand κατόπιν ζητήσεως και αυτό είναι μια επιθυμία που διατύπωσε και η Επιτροπή Προπολογισμού. Θα πρέπει βέβαια όταν μιλάμε για διερμηνείς να ξέρουμε ότι εγκαίρως πρέπει να γνωρίζουμε πόσους εξωτερικούς διερμηνείς χρειαζόμαστε οι οποίοι προσλαμβάνονται ενδεχομένω ένα χρόνο πριν και στο, την τελευταία στιγμή κάνουμε μικροπροσαρμογές. Βραχυπρόθεσμα μπορούμε να κάνουμε κάτι, όχι όμως πολλά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να διερευνήσουμε καλύτερα πόσο θα εργαστούμε περισσότερο on demand και να μην προσφέρουμε υπηρεσίες οι οποίες δεν χρειάζονται για για τους ευρωβουλευτές. Η κυρία Χολμάιγερ αναφέρθηκε στο γραφείο ταξιδίων ε, εσωτερικά ή εξωτερικά τι είναι ακριβότερο. Έχουν γίνει γραπτός ορισμένες ε, ε, παρατηρήσεις διότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες business, τρεις κατηγορίες economy. Αυτό που είναι καλό να γνωρίζουμε είναι ότι το γραφείο ταξιδίων δεν κερδίζει αν υπάρχουν υψηλότερες τιμές διότι τότε μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι το κέρδος τους υποκινεί. Αυτό όμως δεν ισχύει. Όσον αφορά τους οδηγούς θα απευθυνθούμε στο Προεδρείο με μία πρόταση αναμορφώσεως του υπηρεσίας οδηγών. Σε άλλες περιπτώσεις έχω πει ότι μπορούμε να έχουμε όφελος για εσωτερικά εσωτερικές υπηρεσίες ε, για ασφάλεια και ε, για άλλους λόγους αλλά πιστεύω ότι για τους οδηγούς καλύτερα είναι η υπεργολαβία διότι ιδίω αργά το βράδυ καλύτερο είναι να μπορούμε να μην χρειαστεί να επικαλεστεί κανείς το καταστατικό να υπάρχει ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα αποδώσει περισσότερο από ότι υπάρχει Ελπίζω ότι έχω απαντήσει τουλάχιστον στις βασικές ερωτήσεις. Θα επανέλθω στον κύριο Σόρεγκαρντ ε, μεταξύ μας ε, για να του διευκρινίσω ορισμένα θέματα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο, για τον επόμενο χρόνο λοιπόν θα σας υποδείξουμε ως παράδειγμα για το προς μίμηση, προς το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για δεύτερη φορά φέτος, το εκτιμούμε ιδιαίτερος και πιστεύω πως έτσι ολοκληρώσαμε και την εξέταση του σημείου 8 της ημερήσιας διάταξης. Στο σημείο νέα στα διάφορα δεν έχω κάτι να σας ανακοινώσω και 10 είναι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης που θα είναι 10 Νοεμβρίου. 5η ε, με συγχωρείτε 10 Νοεμβρίου όπου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα μας υποβάλει την αιτήσια του έκθεση. Σας ευχαριστώ. Πέρα της συνεδρίαση.